Bien, chers Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. have Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε τη συνεδρίασή μας, γιατί μετά θα πρέπει να ζητήσουμε από του διερμηνείς να μείνουν παραπάνω και δεν το θέλω αυτό, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, επί τη ημερησίας διατάξεως. Θα έχετε ενημερωθεί, συνάδελφοι, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα θυμόσαστε ότι το ζήτησαν οι συντονιστέ, και γι' αυτό ε, ρωτήσαμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν γίνεται μετά από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αν υπάρχει δυνατότητα να συμπεριλάβουμε στα κείμενά μας ε, ποσά στη νομική βάση. Γιατί στην έκθεση της κυρίας Κοστέλο βρισκόμαστε σε αυτό το παράδοξο. Δηλαδή όλες οι επιτροπές που θα γνωμοδοτήσουν ε, ψηφίζουν ε, νούμερα και εμείς είμαστε η μόνη επιτροπή που δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε, να είναι γνωστά πια τα νούμερα, τα ποσά. Ο πρόεδρος λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας ε, απάντησε ως εξής. Μας ζήτησε να αναβάλουμε την ψηφοφορία γιατί αυτή τη βδομάδα λαμβάνει η χώρα ένας τριμερής ε, διάλογος σε πολύ υψηλό επίπεδο, πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και το θέμα αυτό της σύνδεσης των ποσών του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου με την νομική βάση θα συζητηθεί ακριβώς. Αυτό λοιπόν επιθυμεί ο πρόεδρος, συνεπώς και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να αναβάλουμε την ψηφοφορία για τις 20 Μαΐου, στο Στρασβούργο δηλαδή θα ψηφίσουμε. Στις 7 καταφέραμε και πετύχαμε αυτή την ώρα. Βέβαια σήμερα θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων για το πώς έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά την έκθεση αυτή της κυρίας Κοστέλιο. Και θα εξετάσουμε και τις συμβαστικές τροπολογίες. Κατά τα άλλα, όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Ντόιτς. Εδώ δεν χρειάζεται να εξετάσουμε τις συμβαστικέ τροπολογίες, μια που έχει αποσυρθεί το σημείο αυτό από την ημερήσια διάταξη. Και συνεπώς η ανταλλαγή απόψεων για τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα εξεταστεί αμέσως μετά τις ψηφοφορίες, δηλαδή μετά το σημείο 6, λέει ο Πρόεδρος. Το έχει ζητήσει, φαντάζομαι, η συγκήτρια. Εντάξει, συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη. Καλώς, εγκρίνεται λοιπόν. Ανακοινώσεις της Πρόεδρου. Είναι πια παράδοση. Πρώτον, ότι η διερμηνία η οποία δεν χρησιμοποιείται κατά τον τριμερή διάλογο για την ε, ευθύνη της, του κράτους ε, σημαία. εκεί υπάρχουν γαλλικά και αγγλικά, αυτά έχουν ζητηθεί για δύο ευρωβουλευτές. Ο κύριος Τσαμπόρη και ο κύριος ε, Πατρίκ Λιγιάρικο. Δεν συμμετείχαν όμως στην συνεδρίαση αυτή, δεν ενημέρωσαν εκ των προτέρων τη γραμματεία Οπότε, εφ' εξής, ο τριμερής αυτός διάλογος θα γίνεται μόνο στα αγγλικά. Γιατί δεν παρευρέθηκαν που ζήτησαν διερμηνία στις γλώσσες τους. Επίσης, να σας πω ότι η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Σημείο 3 τώρα. Έχουμε να εξετάσουμε τις τροπολογίες στην πρόταση για προφορική ερώτηση όσον αφορά το σύμφωνο δεσμη πιο σωστά για κοινωνικές επενδύσεις. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εγγράφεται στα πλαίσια μιας γενικότερης στρατηγικής αλλά και στα πλαίσια της χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου υπέρ κοινωνικών επενδύσεων. Υπάρχουν 145 τροπολογίες, έχουν κατατεθεί 145 τροπολογίες, 9 έχουν να κάνουν με την προφορική ερώτηση, αλλά εδώ χρειάστηκε Σήμερα βέβαια πρέπει να το αποφασίσουμε. Την έγκαιρη κατάθεση. Για τις 145 τώρα τροπολογίες. Ας δούμε πρώτα την προφορική ερώτηση αυτή καθε αυτή. Εδώ σας είπα έχουμε εννέα τροπολογίες. Τροπολογία αριθμός 1, Καρνόχ, που προτείνει να περιορίσουμε το θέμα της κρίσης, το θέμα της δημοσιονομικής κρίσης της ζώνης ευρώ. Η κρίση βέβαια είναι ευρύτερη από αυτό. Οπότε εγώ προτείνω να μην στηρίξουμε αυτή την τροπολογία. Στη συνέχεια υπάρχει η τροπολογία DeBacker που θέλει να τροποποιήσουμε στην πρώτη ερώτηση τον όρο «enhance» Όχι, in λέει τώρα ο πρόεδρος. όσον αφορά τη στρατηγική μας για το Ευρωπαϊκό Εξάμενο. Ο κύριος Δεβάκερ προτείνει λοιπόν μία τροπολογία εδώ, προκειμένου να μειώσουμε κάπως, να βλύνουμε κάπως την τροπολογία αυτή και απλώς να βάλουμε να ληφθεί υπόψη. Taking in account. Το προτείνω σαν συμβιβασμό. To translate ή to have as a key part. Κάτι το οποίο να μας επιτρέψει να έρθουμε σε ένα συμβιβασμό ανάμεσα στις δύο θέσεις. Ελπίζω να συμφωνήσουμε τελικά. Στη συνέχεια υπάρχει η τροπολογία της κυρίας Λάμπερτ, η οποία επιμένει στη διάρθρωση ανάμεσα στις προτάσεις αυτές και τις συστάσεις σε δημοσιονομικά ζητήματα. Νομίζω ότι μπορούμε αυτό να το προτείνουμε. Έπειτα υπάρχει η τροπολογία του κύριου Ντεμπάκερ πάλι, που προτείνει να διαγράψουμε το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την αναφορά διορθώνει Πρόεδρος του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ζητάει να στηρίξουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πακέτο, τη δέσμη αυτή δηλαδή μέτρων. Η κυρία Λάμπερτ επίσης αναφέρεται στον όρο, στο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, νομίζω ότι είναι ευπρόσδεκτη η τροπολογία της αυτή. Στη συνέχεια, τροπολογία Κάμπρνοχ, πάλι που προτείνει να διαγράψουμε το τρίτο σκέλος της ερώτησης, την τρίτη ερώτηση ουσιαστικά, εγώ νομίζω ότι είχαμε συμφωνήσει να τη διατηρήσουμε. Και υπάρχει και άλλο θέμα, άλλη τροπολογία του κύριου Τεμπάκερ, που αυτή όμω με απασχολεί κάπως. Γιατί προτείνει η ερώτηση 3 να αρχίσει με το εξή. Πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εκπονήσει ένα συγκεκριμένο ρόλο κτλ. Εγώ είχα προτείνει αρχικά να είμαστε υπέρ της τροπολογίας αυτής, αλλά τελικά ως κοινοβούλιο ψηφίσαμε ότι ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει ένα τέτοιο χαρτιπορίας. Οπότε είναι σαν να πηγαίνουμε πίσω με την τροπολογία αυτή. Γι' αυτό και προτείνω να μην τη στηρίξουμε. Για να μην έτσι είναι σαν να προκαταλαμβάνουμε ότι δεν γίνεται αυτό που θέλει το Κοινοβούλιο. Η κυρία Λάμπερτ λοιπόν προτείνει και την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου και τέλος η τροπολογία 9 έχει αποσυρθεί, πρέπει να ξέρετε. Όσον αφορά την πρόταση ψηφίσματο αυτή καθ' αυτή, και τις τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματος, μπορούμε να ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση. Ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς όσους ε, συνέταξαν και υπέβαλαν τροπολογίες. Πολλές θα τις στηρίξω, αλλά προτείνω να συζητήσουμε με τους συντάκτες των τροπολογιών για συμβαστικές τροπολογίες που βεβαίως θα προσπαθήσω να σας υποβάλω αφού προηγουμένως έχω ακούσει βέβαια τα επιχειρήματα των συντακτών των τροπολογιών αυτών που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Γιατί τελικά έχουμε μέχρι τις 30 Μαΐου προκειμένου να εγκρίνουμε το σχέδιο αυτό. Αυτό έχω να σας πω λίγο πολύ ο κύριος Σωρή, μετά ο κύριος Σέρκας, ο κύριος Δεμπάκερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να πω. Δεν ε, έχουμε στείλει τροπολογίες ε, για την ε, προφορική ερώτηση, αλλά γενικά συμφωνούμε με όσα είπατε και τα υποστηρίζουμε. Θα θέλαμε να ζητήσουμε κάποιες τροπολογίες που αφορούν την διατύπωση ή γλωσσικού χαρακτήρα. Αλλά γενικότερα σα υποστηρίζουμε, Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σέρκα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Από τη Σοσιαλιστική Ομάδα πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που προσπαθεί να καλύψει στόχους για την ευημερία και την, την της και των πολιτικών των κοινωνικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά συμφωνούμε με τα όσα είπατε για τις εννέα τροπολογίες που παρουσιάστηκαν και θα ψηφίσουμε έτσι όπως προτείνατε και για το ψήφισμα έχουμε παρουσιάσει διάφορες τροπολογίες γιατί τι θέλουμε πριν από το Συμβούλιο του Ιουνίου να παρουσιάσουμε θέσεις που έχουν ε, επικυρωθεί από αυτή την Επιτροπή και θέλουμε να έχουμε ένα σύνολο μέσων ευρωπαϊκής ε, διακυβέρνησης. Θέλουμε να έχουμε δείκτες κοινωνικούς, θέλουμε να ληφθεί υπόψη στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο οι κοινωνικές επενδύσεις να ληφθούν υπόψη και θέλουμε να αναγνωριστεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των Συμβάσεων της ε, ΟΕ. Επίσης θέλουμε μια αναφορά στην αναγκαιότητα να υπάρχει επένδυση σε κοινωνικές κατοικίες στην Ευρώπη καθώς ε, έχουμε κρίση στα κίνητα σε πάρα πολλές χώρες, το δούμε των κινητών σε πολλές χώρες και επίσης ε, θα θέλαμε να συμπεριληφθούν κάποιες τροπολογίες που αφορούν περισσότερο το θεωρητικό τμήμα της ανακοίνωσης της Επιτροπής όπου Υπάρχει κάτι με το οποίο συμφωνούμε, αλλά ε, θα μπορούσαμε να δεχθούμε σε σύγχυση ε, και θα θέλαμε να ξεκαθαριστεί ότι οι παραδοσιακές λειτουργίες της κοινωνικής πρόνοιας, ε, δηλαδή της πολιτικής του κράτους πρόνοιας, θα χρησιμοποιηθούν και θα συμπληρωθούν, και θα με τις δύο νέες λειτουργίες ε, που ε, έχουν εισαχθεί στο γενετικό μας κώδικα στην εποχή της κρίσης ε, και είναι η επένδυση και η σταθεροποίηση της οικονομίας. Πρόκειται για δύο λειτουργίες που αναμφισβήτητα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το σύστημα κοινωνικής πρόνοια, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για προστασία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι ευάλωτοι, ηλικιωμένοι, άρρωστοι και πρέπει να προστατεύονται γιατί δεν μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες. Ε, όλο ένα και περισσότερο ε, απλώς ε, θεωρούμε ότι είναι η οικονομική αυτή η φορής ε, κοινωνικής προστασίας. Όμως ε, είδατε ότι η κρίση είναι πάρα πολύ σκληρή και θα πρέπει αυτοί οι φορείς να χρησιμοποιηθούν ε, ε, όχι μόνο ως ε, φορείς κοινωνικών επενδύσεων, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για κοινωνική προστασία, γιατί δεν είναι όλοι σε θέση να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και αυτό μπορεί να συμβαίνει και για βιολογικούς λόγους, όχι μόνο για λόγους οικονομίας της αγοράς. Ευχαριστώ κύριε Στυμπάκερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα ήδη ανέφερα στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων ότι υπάρχει ισορροπία τόσο όσον αφορά το σχέδιο του ψηφίσματος όσο και την ερώτησή σας. Οι δικές μητροπολογίες έχουν ως στόχο να διευκρινίσουν τα θέματα τα οποία θέλουμε να θέσουμε στην Κομισιόν. Παραδείγματο χάρη όσον αφορά την πρώτη σας πρόταση ε, για τη χρήση της λέξης μετάφραση. Αυτό είναι αποδεκτό για μένα. Ε, κατά τα άλλα, όσον αφορά τις άλλες ε, τροπολογίες για το σχέδιο του ψηφίσματος, ε, ε, νομίζω ότι δεν πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Η έκθεση είναι αρκετά ισορροπημένη. Ορισμένα από τα στοιχεία που είναι σημαντικά για μας, ε, για την ομάδα μας, είναι ότι πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στον εξυγχρονισμό του συστήματος πρόνοιας. Και επίσης τα εργαλεία που υπάρχουν να εκλειφθούν ως κίνητρα από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Η θέση απασχόλησης είναι καλύτερη προστασία από την φτώχεια. Επίσης, οι τροπολογίες μας επιθυμούν να διευκρινίσουν την βιωσιμότητα των κοινωνικών δαπανών, όπως και την σωστή χρήση νέων εργαλείων, έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα στους πολίτες. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας κοινός στόχος όλων μας. Έτσι λοιπόν οι τροπολογίες μας κατατέθηκαν ε, σε αυτό το πνεύμα και ελπίζω να συζητηθούν κατά τη διάρκεια των ε, συζητήσεών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. να δώσουμε το ρόλο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν και να κάνω και μία παρατήρηση στο παράδοπο σε λίγες Κάποιος ακόμη ζητά το λόγο. αλλά να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω. Για τον τίτλο ήθελα να πω κάτι, δεν το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Γιατί μιλάμε για ένα σύμφωνο κοινωνικών επενδύσεων. Πρόκειται για ένα πακέτο που έχει πολλούς πυλώνες, για μια δεσμή μέτρων που έχει πολλούς πυλώνες. αλλά δεν καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά αν μιλάμε για το κοινωνικό σύμφωνο επενδύσεων, αν ε, μιλάμε για την ε, χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τομείου. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον τίτλο της ανακοίνωσης, αλλά ε, εγώ νομίζω ότι είναι κάπως ατυχής και δεν μας διευκολύνει να καταλάβουμε ακριβώς τι λέει το κείμενο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα και στο παρελθόν, υποστηρίζω αυτή την έκθεση. Μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντική. Κάποιες τροπολογίες που έχω καταθέσει, θέλω να υπογραμμίσω. Αναφέρομαι και στα κοινωνικά δικαιώματα των μεταναστών, που είναι σημαντικό επίση. Είναι σημαντικό κινητικότητα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να λαμβάνει χώρα και επίσης είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ε, και σε αυτό αναφέρεται η τροπολογία μου. Και επίσης ένα συνδέσμος που φαίνεται πολύ σημαντικός είναι ο συνδέσμος μεταξύ της ενίσχυσης κοινωνικών δικαιωμάτων και του θέματος της υποστήριξης ε, των ε, εταιριών κοινωνικής οικονομίας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, όσον ε, αφορά στο σχόλιο σας ε, ότι το πακέτο είναι μεγάλο, ότι περιλαμβάνει διάφορα έγγραφα όσον αφορά τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει εμπνευστεί από το πακέτο της απασχόλησης. Θελήσαμε να καταθέσουμε ένα περιεκτικό πακέτο που να αφορά και στη διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, η οποία δεν μπορεί να αφορά ένα και μόνο έγγραφο το οποίο να ε, επιλαμβάνεται του κράτους πρόνοιας και των κοινωνικών επενδύσεων. Εμείς θελήσαμε τις ε, κοινωνικές επενδύσεις να τις εξετάσουμε κάτω από ένα ευρύτερο πρίσμα. Γι' αυτό λοιπόν ε, θελήσαμε να δώσουμε και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η Κομισιόν θέλω να σας πω ότι εγκρίνει και επαυξάνει όσον αφορά αυτά που λέτε για το πακέτο και στηρίζει τις δικές σας τις προτάσεις, ε, κυρίως ε, όσον αφορά στην αντιμετώπιση της ενεργείας για τους νέους, ε, πρέπει να δούμε ότι ε, πράγματι πρέπει να επιτευχθεί κάποια ισορροπία. Πολύ χρήσιμα όλα αυτά που θίξατε και αυτά βέβαια αναφέρονται στα έγγραφα που έχουν κατατεθεί και στην ανακοίνωση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές ε, κοινωνικές ε, προκλήσεις και η Κομισιόν καταλήγει στην άποψη ότι χρειαζόμαστε μια περιεκτική προσέγγιση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό εξηγείται αυτή, αυτός ο όγκος του πακέτου, το, το πακέτο είναι μεγάλο. Σας ευχαριστώ πολύ για όσα είπατε όσον αφορά τις τροπολογίες. Ευχαριστώ τον κύριο Ρή για την στήριξή του, τον κύριο Σερκάς. Εντάξει, το φαντάζεστε ότι θα σας χρειαστώ για τις συμβαστικές προτάσεις. Με τον κύριο Ντεμπάκερ έτσι κι έχουμε τη συνήθεια να συνεργαζόμαστε, οπότε φαντάζομαι ότι θα καταλήξουμε, σε, ελπίζω τουλάχιστον, θα καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις μαζί όσο και αυτό που είπε η κυρία Μπεναράτου, αυτά είναι θέματα τα οποία ε, πιστεύω ότι είναι σωστά απριόρι. Και σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε στο θέμα του συντονισμού των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης, όπως επίσης και στους μετανάστες, που στο αρχικό κείμενο δεν συμπεριλαμβάνονται, αλλά θα πρέπει. Οπότε θα επανέλθω με μια πρόταση πάνω σε αυτά τα σημεία που ελπίζω να στηριχθεί όσο γίνεται περισσότερο. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες στις 29 Μαΐου και να ψηφίσουμε στις 30 Μαΐου. Στην Ολομέλεια θα πάει το θέμα τον Ιούνιο στο Στρασβούργο, 10 με 13 Ιουνίου δηλαδή. Σημείο 4. Το έχουμε αναβάλει. Οπότε, περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε πρώτα το κείμενο της προφορικής ερώτησης. Σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς ε, κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή. Εφαρμογή των ε, μέτρων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 2014-2020, σύμφωνα με τόσα συζητήσαμε. Υπενθυμίζω επίσης στους συναδέρφους ότι για την τροπολογία ρυθμός 2 ο κύριος Ντεμπάκερ δέχτηκε μια προφορική τροποποίηση η οποία έχει σαν αποτέλεσμα το taking in account, να λαμβάνουμε υπόψη, να ε, αντικατασταθεί από το to translate, να μεταφράσει, να ερμηνεύσει. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ της πρώτης τροπολογίας, Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία τώρα, η δεύτερη με την τροποποίηση υπέρ. Σέρκα, μην ψηφίζεις κατά, είσαι υπέρ. Με την προφορική τροποποίηση είσαι υπέρ λέει η πρόεδρος. Υπέρ λοιπόν. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 της Jean Lambert υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ερώτηση 2. Τροπολογία 4 του Φιλίπ Ντεμπάκερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5, Τζιν Λάμπερτ, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Μίλαν Κάμπνοχ, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8, Τζιν Λάμπερτ, υπέρ. Κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 7, Φιλίπ Ντεμπάκερ. Είναι κατά η συγκήτρια. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 9 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε λοιπόν το σύνολο του κειμένου τώρα. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. 36 υπέρ, μία ψήφος κατά και καμία αποχή. Εγκρίνεται. Σχέδιο γνωμοδότηση του συναδέλφου μας Ταμάς Ντόιτς. Πρόκειται για γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη μια βιοοικονομία για την Ευρώπη. Αυτό είναι ο τίτλος. Έχουμε τρεις τροπολογίες συμβαστικές, τρεις συμβαστικές. Θέλετε το λόγο? Παρακαλώ κύριο Ρή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει κάποιο λάθος στον κατάλογο ψηφοφορίας του ΕΛΚ όσον αφορά την τροπολογία αριθμός 12 Αντί για μείον πρέπει να έχουμε συν. Είναι για το έλκα αυτό που το λέω. Καλώς. Εντάξει, βοηθάμε έτσι το ΕΛΚ να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Ψηφίζουμε παράγραφος τροπολογία 6, σαρία σαγιά. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την πρώτη παράγραφο, με τροπολογία 7 της Αντιγόνης Παπαδοπούλου υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 1, πάντα έχουμε την τροπολογία 8 της Αντιγόνης Παπαδοπούλου και του Αλεχάνδρου Θέρκας, που ψηφίζουμε κατά δύο τμήματα, αλλά το δεύτερο τμήμα έχει αποσυρθεί, οπότε ψηφίζουμε μόνο το πρώτο τμήμα. Points out that anticipation μέχρι opportunities in Europe. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 10 σαρίσα για υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 2, τροπολογία 11, Αντιγόνη Παπαδοπούλου. Με ναι, προφορική τροποποίηση. Δεν υπάρχει αντίρρηση για αυτήν. Ωραία, ψηφίζουμε την τροπολογία 11 υπέρ, κατά αποχές Εγκρίνεται. Μετά την παραγραφό 2, τροπολογία 12, Αντιγόνη Παπαδοπούλου. Και το είναι υπέρ, να ξέρετε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3, τροπολογία 13, Φίλιπ Μπενιό. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14, Σερίες Αγιά. Εδώ υπάρχει προφορική τροποποίηση Υπάρχει αντίρρηση για αυτήν. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν τροπολογία 14 τροποποιημένη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Συμβαστική τροπολογία α του ΕΛΚ και των σοσιαλιστών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 της κυρίας Αντιγόνης Παπαδοπούλου. Εδώ θα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4, τροπολογία 16. Πάλι τη Αντιγό Παδοπούλου υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 17, Σαρία ΣΑΓΙΑ Με προφορική τροποποίηση. Δεν έχετε αντίρρηση. Όχι, ψηφίζουμε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 18, υπέρ, κατά. Υπέρ, κατά αποχές θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Το πρώτο ή το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε. Για ξαναπείτε τι ρωτήσατε, δεν σας κατάλαβα, λέει η Πρόεδρος. Ψηφίζουμε το πρώτο ή το δεύτερο. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Πέρα στις ψηφοφορίες. «21 ψήφι υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται». Παράγραφος 6. Συμβαστική Β. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 6, τροπολογία 21, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7, τροπολογία 24, Σάρια Σαγιά, υπέρ, κατά αποχές θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 24. Ψηφίσατε όλοι πέρα της υποφορίας 27 υπέρ, 14 κατά. Εγκρίνεται. Μάλλον δεν είχατε σηκώσει τα χέρια σας στην αρχή. Λοιπόν, τώρα έχουμε τη συμβαστική γάμα. Υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. 25 σαρίσα για υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9, τροπολογία 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10, 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στο υλικό 1, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το Β, έχουμε τροπολογία 2, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3, Παπαδοπούλου υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4, Παπαδοπούλου υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 5, Παπαδοπούλου υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά το σύνολο του κειμένου. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. 40 υπέρ, μία ψήφος κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγητριά μας που δεν τη βλέπω όμως εδώ. Ολοκληρώσαμε με τις ψηφοφορίες. Πολύ σύντομη ήταν ε, σήμερα η διαδικασία αυτή και να περάσουμε στο σημείο 10 όπου θα δώσω το λόγο στην συγγήτρια, την κυρία Μόριν Σαρτιέ, για να μας ε, παρουσιάσει την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο στο πλαίσιο του 15ου και 16ου Τριμμένου Διαλόγου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το σημείο αυτό. Χθες το βράδυ υλοποίησαμε το 16ο τριμερ διάλογο για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και προσεγγίσαμε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Nous abordions hier συζητήσαμε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα χθε το βράδυ. Σα παρακαλώ, δεν είναι δυνατόν να γίνονται συζητήσει. και κλεισμένο το θαχτηρών σχεδόν συμβαίνουν οι τριμερεί διάλογοι και εδώ πρέπει να το δημοσίσουμε. Μιλάμε για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Έτσι λοιπόν σα παρακαλώ να ενδιαφέρεστε να αποχωρήσετε από την αίθουσα και να επιτρέψετε στην εισηγήτρια να μας ενημερώσει υπό τι βέλτιστε συνθήκε. Μάλιστα, ευχαριστώ λέει η Χθε το βράδυ, λοιπόν, υλοποιήσαμε το 16ο τριμερή διάλογο για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ο χθεσινό ε, τριμερή διάλογο επικεντρώθηκε στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και τη σχέση με την εγγύηση για τους νέους. Πιστεύω ότι το πρώτο σημείο επί το οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε είναι το εξή. Να ξέρουμε ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είναι για την Επιτροπή ένα γενές μέρος της εγγύσης για τους νέους, αλλά κατόπιν συζητήσεως διαπιστώνουμε ότι από την πλευρά του Συμβουλίου δεν ε, βλέπει το Συμβούλιο με τον ίδιο τρόπο την διάρθρωση μεταξύ της εγγύησης για τους νέους και της πρωτοβουλίας για την ε, απασχόληση των νέων. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πρώτο πρόβλημα που είναι πρόβλημα σύλληψης ε, της εγγύησης για τους νέους και ποια είναι η σχέση της σε σχέση με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Να σας πω ότι εδώ φαίνεται ένα δικαίωμα για ό,τι σκεφτόμουν πάντα ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ε, δεν αποτελεί παρά μια πολιτική απόφαση με μια πολιτική παρουσίαση και αυτή αποτελεί ένα μέρος της ουσιαστικής ε, δουλειάς ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει για πρώτο στόχο να μπορέσει να βοηθήσει τους ε, νέους ε, να βρουν απασχόληση και τους νέους με προσόντα να μπουν στην αγορά εργασίας κατελήλως. Χτες ε, το βράδυ, λοιπόν, επειδή όλα αυτά δεν είναι ξεκάθαρα, ρωτήσαμε το Συμβούλιο να μας πει ποιο θεωρεί ότι είναι η διαφορά των πολιτικών στόχων και των στόχων ε, σε ό,τι αφορά την ανάληψη δράσης ε, μεταξύ των δύο, μεταξύ της εγγύσης και της πρωτοβουλίας. Η δική μας ερώτηση απλά επιζητούσε στο να υπάρχει μια πολιτική διευκρίνηση, αλλά δεν λάβαμε απάντηση, γιατί το Συμβούλιο μας είπε ότι δεν είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν, εξακολουθεί να παραμένει αυτό το ερωτηματικό αλλά εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα και παραμένει εκρεμές. Το δεύτερο σημείο το οποίο συζητήσαμε είναι ε, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, δηλαδή για την ε, ηλικική ομάδα. Ξέρετε ότι στο κοινοβόλιο η δική μας ψηφοφορία ήταν ε, σαφής, γιατί εμείς θέλαμε αυτή η πολιτική απόφαση για την ε, πρωτοβουλία, για την επασχόληση των νέων, ε, όχι μόνο να καλύπτει, όχι μόνο ε, τους ε, νέους 15 με 24, 15-24 ετών, αλλά και τους νέους πτυχιούχους, οι οποίοι μπορεί να συνεχίζουν μάλιστα τις σπουδές τους, αλλά είναι άνεργοι. Και βλέπουμε τι συμβαίνει σε μια χώρα όπως η Ισπανία, πόσοι ε, τέτοιοι νέοι πτυχιούχοι υπάρχουν και είναι άνεργοι και μπορούν, θα μπορούσαν να αποφεληθούν από μια εγγύηση, από μια τέτοια πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αν περάσουμε από την ηλικία 15-24 στην ε, ε, στην στην και ομάδα 15 30 οτών. και τότε δούμε ότι πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των δικαιούχων, τότε θα φανεί ότι θα έχουμε μια πραγματική πολιτική για τους νέους που θα καλύπτει και την περίοδο ένταξης στην αγορά εργασίας μέχρι τα 30 έτη. Εκεί θα έχει η δική μας ψήφος πραγματικό πολιτικό νόημα. Η δική μου εντύπωση είναι τα έξι ε, δισεκατομμύρια που είναι τρία συν τρία δεν καλύπτουν παρά ένα πολύ μικρό ποσοστό των αναγκών. και νομίζω ότι πραγματικά έχουμε μία πολύ μεγάλη μάχη μπροστά μας. Τρίτο σημείο, Πρόεδρε, αφορά τη θεματική συγκέντρωση. Η θεματική συγκέντρωση θα συμπεριλαμβάνει και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ή όχι. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Ούτε και εδώ είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος σχήματο. Δεν θυμάστε ότι στη θεματική συγκέντρωση η πρόταση της Κομισιόν είναι να επικεντρωθεί σε τέσσερις σημαντικούς άξονες να συγκεντρώσει τέσσερι τέσσερις άξονες τις ε, πολιτικές των κρατών μελών, ενώ εμείς ε, θα θέλαμε να είχαμε ε, έξι, επτά άξονες, ίσως μεσοπρόθεσμα, να προτείναμε. Αυτή η πολιτική απόφαση πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων να μπορούσε να προσθεθεί στη συγκέντρωση τεσσάρων προτεραιοτήτων ή να αποτελέσει εγγενές τμήμα των έξι που ζητάμε. Θα δούμε εδώ λοιπόν πώς θα διαπραγματευτούμε. Αυτή είναι είναι αποτελεσει εγγενες τμημα των εξι που ζηταμε θα δουμε εδω λοιπον πως θα διαπραγματευτουμε αυτη ειναι η συνοψη των όσων ε, προβλημάτων συζητήσαμε χθε το βράδυ, αλλά αν μου επιτρέπετε και ένα προσωπικό σχόλιο για το χθεσινό τριμερή διάλογο, συνειδητοποιούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ήταν ε, μια απόφαση που παρουσιάστηκε πάρα πολύ γρήγορα, όμως ε, σήμερα στα θέματα ουσίας ακόμα δεν έχουμε λάβει απαντήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. ο κύριος Σέρκας. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω μήπως θα ήταν χρήσιμο σε αυτό το στάδιο να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρώτο τουλάχιστον σημείο που χρειάζεται διευκρινήσεις νομίζω. Η πρωτοβουλία έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσως θα ήταν καλό. Μήπως λοιπόν να ακούσουμε πρώτα την Επιτροπή ή θα αρχίσουμε τώρα τον γύρο των παρεμβάσεων των Ευρωβουλευτών δηλαδή. Δεν θα μας εξηγήσει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ θα ήθελα να μου διευκρινίσουν πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Είμαστε λοιπόν εν μέσω πλήρης σύγχυσης και μπερδέματος. Προληπτικά λοιπόν θα ήθελα να μεταφέρουμε στην Επιτροπή και το Συμβούλιο το εξής. Εμείς ξεκινήσαμε με την πρωτοβουλία για τους νέους και ζητήσαμε μια ευρωπαϊκή εγγύηση. Ενώ τώρα καταλήγει να είναι κάτι που πρέπει να στηρίξουν οι χώρες μέλη. Εμείς θέλαμε να είναι μια πραγματική πολιτική και όχι μόνο στα λόγια. Να μην μείνει μία από τις πολλές υποσχέσεις που έχουμε κάνει προς τους Ευρωπαίους πολίτες και οι οποίοι τελικά βλέπουν ότι μεταφέρονται στις ελληνικές καλένδες, ότι δεν υλοποιούνται ποτέ. Δεν θέλουμε λοιπόν να είναι μια ακόμα υπόσχεση ενώ πρόκειται για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα για τους νέους. Δεν είναι δυνατόν όμως να παραμένει η σύγχυση. Έχουν περάσει τρεις μήνες και όταν διάφοροι πρωθυπουργοί και καγκελάροι λένε ότι τον Ιούνιο και ο Ισπανός πρωθυπουργός και ο Ιταλός είπανε ότι τον Ιούνιο αυτό θα γίνει. Θα... Δεν βλέπω πώς είναι δυνατόν το Συμβούλιο να λέει ότι δεν έχει να πει τίποτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ούτε μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ερμηνεύει την απάντηση του Συμβουλίου. Πάντως άκουσα την Ελίσαμπετ και θέλω από πλευρά της ομάδας μου να στηρίξω, γιατί πιστεύω ότι η μάχη που δίνει είναι σωστή και δίκαια. Το πρόγραμμα τελικά είναι για τους μισούς νέους ή για όλους. Ποσοτικά δηλαδή αναφέρθηκε στους διπλωματούχους. Οπότε τελικά θα είναι μια πρωτοβουλία για τους μισούς Ευρωπαίους νέους ή για όλους. Στην ίδια λογική λοιπόν λέω ότι θα πρέπει να είναι μια πραγματική δέσμευση και όχι μόνο λόγια και πρέπει να αγωνιστούμε μέχρι το τέλος, ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι νέοι που έχουν ένα πρόβλημα ένταξης στην αγορά εργασίας να μπορέσουν είτε έχουν δίπλωμα είτε δεν έχουν δίπλωμα να αποφεληθούν από ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τέλος, για την θεματική συγκέντρωση. Είναι ξεκάθαρο ότι αν το Συμβούλιο τον Ιούνιο έχει το θέμα των νέων σαν κύριο άξονα, θα είναι πολύ καλό οι δικές μας οι πολιτικές να είναι συνεκτικές μεταξύ τους και να μην επικρατεί χάος και μπέρδεμα που θυμίζει μια τρέλα. Ο κύριος Μάν, Τόμας Μάν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά την ε, Ελίζαμπετ. Γιατί... Είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε εδώ. Κοιτάξτε, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ καλή η δουλειά σου. Ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε. Ε, χρειαζόμαστε ε, δεσμευμένους και στρατευμένους συνεργάτες. Αυτό που είπε και πίσω ο Αλεξάνδρο, δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν μόνο τα στοιχεία, πρέπει να υπάρχει και αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε δηλαδή να συνεχίσουμε απλά να καταγράφουμε ότι η ενεργεια των νέων σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι τόσο υψηλή που ορισμένοι να έχουν την εντύπωση, οι νέοι δηλαδή, ότι γεννήθηκαν σε λάθος ε, χρονική στιγμή. Δεν μπορούμε να τα δεχόμαστε αυτά. Ξέρετε, εγώ έρχομαι από μια τέτοια χώρα και τη λίστη βρήκαμε από κοινού. Οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι, οι κοινωνικοί εταίροι. Πρέπει βέβαια να υπάρχει και το σωστό πολιτικό πλαίσιο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι με την εγγύηση για τους νέους με αυτή την πρωτοβουλία δεν πρέπει να οδηγήσουμε σε σύγκρουση, αλλά να λειτουργήσουμε συμπληρωματικά και να πούμε ότι αυτή είναι τομεί ε, στους οποίους πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Το θέμα λοιπόν της ε, ανεργίας δεν μπορεί να σταματάει εκεί όπου θα λέμε ξέρετε υπάρχει οξύ διαχωρισμός. Δεν είναι αυτό, υπάρχουν κοινά στοιχεία, ε, υπάρχουν διαφορετικές εμπειρίες και ορισμένοι έχουν πραγματικά πολύ καλά πτυχία, αλλά και αυτοί πλήττονται από την ανεργία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχουν οι σωστέ πρωτοβουλίε. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Γνωρίζω ότι πολλοί είναι επιφυλακτικοί επ' αυτού. Ξέρω ότι το ίδιο ίσχυσε στην αρχή για το Ταμείο τη παγκοσμιοποίηση και εγώ στην αρχή το επέκρινα, αλλά πραγματικά επέφερε πολλά και θετικά. Και κυρία Πρόεδρε, με το Ευρωπαϊκό, με το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση, με συγχωρείτε, μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Ε, και έτσι λοιπόν ε, υπάρχει το εξή ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλές φορές υπάρχει διάσταση απόψεων, αλλά για αυτό το θέμα χρειαζόμαστε την Επιτροπή με, την, με το μέρος μας. Ελίζαμπεθ, ε, θέλω να σας ρωτήσω, στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο υπάρχει μία περίπτωση όπου να μπορεί κανείς ε, να διαφοροποιήσει ανάμεσα σε βόρεια και νότια κράτη ή μήπως το Συμβούλιο έχει ε, γενικευμένη θέση. Αυτό είναι ενδιαφέρον να το γνωρίζει κανείς. Γνωρίζω ότι ορισμένοι δεν θέλουν να διαραίουν ε, πληροφορίες, θέλουν τις διαπραγματεύσεις και κλεισμένων των θυρών. Εμείς όμως είμαστε διαφανείς. Μεταδίδονται τηλεοπτικά οι συνεδριάσεις μας και έτσι μπορούμε να ελέγξουμε και τα κράτη-μέλη και υποστήριξη μπορούμε να προσφέρουμε μόνο όταν γνωρίζουμε ποιος έπαιξε με τι χαρτιά και πώς. Ελίζαμπετ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν σας δώσω το λόγο στην Καρή ο Αλέξανδρος Θέρκας ε, ρώτησε αν μπορούμε να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι ο στόχος δεν είναι αυτός. Αυτό το κάνουμε στον τριμερή διάλογο. Εδώ αυτό που κάνουμε είναι ότι μεταφέρουμε τόσο συζητήθηκαν στον τριμερή διάλογο εδώ. Δεν μεταφέρουμε δηλαδή τον ίδιο τον τριμερή διάλογο εδώ, απλώς ενημερώνουμε. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να σας κάνουμε να δουλέψετε, αλλά αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ. <clears throat> Μεταφέρουμε, ενημερώνουμε δηλαδή τους ευρωβουλευτές για το όσα έγιναν ήδη στον τριμερή διάλογο. Κάνε μαντελή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και χρόνια ακούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να ασχοληθεί με τους νέους και ότι οι νέοι πρέπει να είναι η προτερότητά της. Οι νέοι όμως είναι τα πρώτα θύματα της κρίσης. Και όσο περνά ο καιρός, τόσο περισσότερο η κρίση αυτή αποδεικνύεται δύσκολη και όλο και περισσότερο οι νέοι βρίσκονται σε δυσκολίες. Όσο περνά ο καιρός, όλο και περισσότερο. Θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι νέοι δεν σας ξεχνάμε. Σύμφωνοι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και συμφωνώ, έχουμε δίκιο που θέλουμε να διευρύνουμε το στόχο αυτό από τα 15 στα 30 χρόνια. Γιατί οι σπουδές κρατάνε όλο και περισσότερο σήμερα. Και τελικά όταν τελειώνει κανείς τις σπουδές του, τότε μπαίνει στις δυσκολίες ως νέος. Όμως, με 6 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Όλοι λένε ότι είναι προτερότητα οι νέοι, ε λοιπόν εκεί βάλτε τα λεφτά. Γιατί το μέλλον της Ευρώπης είναι ακριβώς η νεολαία. Τι λέει το η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Λέει ότι χρειάζονται 21 δισεκατομμύρια ευρώ για να υπάρξει μια πραγματική λύση σε 7,5 εκατομμύρια νέους άνεργους χωρίς προσόντα, χωρίς κατάρτιση. Ενώ το κόστος της αδράνειας, αν δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα, αυτό στοιχίζει 153 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή τι λέμε με τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, εδώ ε, τσακωνόμαστε για ψίχουλα και λυπάμαι που το λέω έτσι, ενώ η πρόκληση είναι τόσο μεγάλη που αν δεν αλλάξουμε ρότα τώρα πάμε κατευθείαν στην καταστροφή. Συνεπώς, στις διαπραγματεύσεις ένα ισχυρό επιχείρημα είναι ότι τα 6 δισεκατομμύρια δεν φτάνουν. Τώρα υπάρχουν 3 δισεκατομμύρια στο κοινωνικό ταμείο και άλλα 3 αλλού. Η θέλησή μας λοιπόν είναι να πιέσουμε προς τον ε, δημοσιονομικό αυτό στόχο και μετά θα δούμε πώς θα τον εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Σήμερα υπάρχει μια σάφια για την υποχρέωση αυτή εφαρμογής του μέτρου από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την ενεργοποίησή της, για την κινητοποίησή της. Σε υλοποιείτε την εντολή που σας δώσαμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ε, τώρα, Επιμένετε από των τριών σημείων. Εγώ χαίρομαι που εμείς έχουμε ανοίξει αυτό το θέμα των 30 ετών, γιατί νομίζω ότι βλέπουμε κάτι που οι άλλοι δεν βλέπουν ακόμη. Μερικές φορές δηλαδή έχουμε δίκιο πολύ νωρίς δυστυχώς ε, και πρέπει να διαφωτίσουμε και τη σκέψη των υπολοιπών. Όμως έχουμε αυτό το στερεότυπο, πιστεύουμε ότι νέοι είναι ως 24 ετών και ακούσαμε το Συμβούλιο να μας λέει όχι, οι πραγματικοί νέοι πρέπει να βοηθήσουμε είναι αυτοί που είναι 15 χρονών. Όμως πραγματικά πρέπει να δώσουμε και μία όθηση για να μην οδηγηθούμε στην καταστροφή γιατί πραγματικά οι άνθρωποι που βρίσκονται σε πραγματικές δυσκολίες είναι αυτοί που είναι από τα 24 στα 30 έτη σε σχέση με το όσα μας περιέγραψε η συγγήτρια και που μας εξέπληξε στο χθεσινό τριμερή διάλογο είναι ο τρόπος ε, με τον οποίο αρνείται το Συμβούλιο να έχει στο κύριο νομοθέτημα οποιαδήποτε αναφορά στην εγγύηση των νέων με ένα νομικό επιχείρημα, όμως μας διαφωτίζει στην ιδέα ότι υπήρχε μια βούληση να κατασκευάσει κάτι που θα μπορούσε να φαίνεται σαν πολιτικό μήνυμα, αλλά χωρίς ε, τελικά να φτάνει μέχρι το τέλος. Και το επιχείρημα είναι ότι δεν θα χρειαζόταν παρά να τεθούν σε εφαρμογή τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη 7ης και 8ης Φεβρουαρίου. Και εδώ η δική μας αντιπροσωπεία είναι πεπισμένη, απόλυτα πεπισμένη ότι όταν ε, δούμε τα συμπεράσματα του Φεβρουαρίου υπάρχει ένα τμήμα που μπορεί άμεσα να αποφασιστεί από το Συμβούλιο και αυτό αφορά τα νούμερα. Εμείς ως Κοινοβούλιο, εμείς μόνο ναι ή όχι μπορούμε να πούμε στο τέλος του όλου εγχειρήματο, αλλά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν μπορεί να προκρίνει την νομοθετική βάση. Εμείς είμαστε συνομοθέτες και είναι η πρώτη φορά που σε τριμερείς ε, διαλόγους συζητούνται τέτοια θέματα. Όμως σήμερα έχουμε μπλοκάρει, έχουμε μπλοκίσει αυτό το σημείο. Δηλαδή αυτό που αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας λένε α, αυτό αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας το λέει το Συμβούλιο όμως εμείς ως νομοθέτης έχουμε δικαίωμα να υψώσουμε τη φωνή μας, να πούμε και αυτό που θέλουμε εμείς. Το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτή την συζήτηση και νομίζω ότι θα πρέπει να ακουστεί αυτό το επιχείρημα γιατί για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ουσιαστικό αυτό το ζήτημα και μάλιστα αν λάβουμε υπόψη ότι σε αυτή την Επιτροπή έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα της εγγύησης των νέων ε, και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να επωφεληθούν μόνο ορισμένες χώρες από αυτά τα εξειδής. Επίσης έχουμε και κάποιες συζητήσεις με την Επιτροπή ε, περιφερειακών υποθέσεων ε, και ξέρετε υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όχι μόνο το θέμα της εγγύσης των, νέων αλλά και για το τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην πολιτική συνοχής. Δεν θα σας αναφέρω τώρα τις λεπτομέρειες των συζητήσεων αλλά εν τέλει από τις 26 ε, Μαρτίου έχουμε ζητήσει τριμερή διάλογο υψηλού επίπεδου που ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί και ε, στον προγραμματισμό μένει αοριστό και μόλις έμαθα ότι η κυρία Χιμνέρ δέχτηκε να έρθει σήμερα το απόγευμα στη συζήτηση στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων. Ε, έτσι λοιπόν, ε, εκ μέρου ε, του Δημικότζα θα σα ενημερώσω. Η κυρία Χίμπνερ μας υπενθυμίζει ότι θέλουμε ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τμήμα να συμμετέχει στο επίπεδο του 25% στην πολιτική συνοχής. Λοιπόν, ο επόμενος τριμερής διάλογος θα λάβει χώρα στις 14 Μαΐου και βεβαίως θα ενημερωθούμε στη συνεδρίαση της 20 Μαΐου. Ε, Σημείο 7α. Σε σχέση με το μη στον των Απόρων. Έχουμε αναβάλει την ψηφοφορία, όπως γνωρίζετε. Αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για τις ε, προτάσεις ε, συμβιβαστικών τροπολογιών και για, για το θέμα αυτό θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Κοστέλο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, αναβλήθηκε για τις 20 Μαΐου η ψηφοφορία. Έτσι έχουμε χρόνο να συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Θέλω να επικεντρωθώ σε τρία ζητήματα σήμερα το πρωί. Το ένα έχει να κάνει με την συμμετοχή στο πρόγραμμα και το δεύτερο είναι ο προπολογισμό και βέβαια το θέμα της πλατφόρμας για τη διάδοση. Όσον αφορά την συμμετοχή, και το πρόγραμμα επισητιστικής βοήθειας. Όπως γνωρίζουν οι ευρωβουλευτές και ιδιαίτερα οι σκιώδεις, αυτό το θέμα για το κατά πόσο συμμετοχή θα είναι σε εθελοντική ή όχι βάση, είναι κάτι που κυριάρχησε τη συζήτηση των σκιωδών για βδομάδες. Στην αρχική έκθεση που υπέβαλα, εγώ δεν υπέβαλα τροπολογίες για το θέμα αυτό της εθελοντικής ή όχι συμμετοχής, γιατί θεώρησα ότι για τους άπορους το σχετικό ταμείο θα έπρεπε να απευθυνθεί σε όλες τις χώρες μέλη και όχι μόνο στις χώρες μέλη που ήταν διατεθειμένες να συμμετάσχουν ή όχι. Τώρα από τις συζητήσεις που έγιναν με τις άλλες πολιτικές ομάδες και πολλές από τις πολιτικές ομάδες σκέφτηκαν ότι είναι καλύτερο να έχουμε ένα σύστημα εθελοντική συμμετοχή στο πρόγραμμα. Καταλήξαμε τώρα σε μια κατάσταση όπου έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες τροπολογιών. Πολλές πολιτικές ομάδες θέλουν τροπολογίες για την εθελοντική συμμετοχή. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν, τότε τα σχετικά κονδύλια μεταφέρονται. Η ομάδα των σοσιαλιστών αποφάσισε ότι πρέπει να μείνουμε στην αρχική μας θέση και ότι το Ταμείο θα πρέπει να απευθύνεται στους άπορους όλες τις χώρες μέλη και ότι θα πρέπει να συμμετέχουν οι χώρες μέλη στην ε, σχετική περίοδο και ότι στο μεταξύ όμως δεν θα γίνει αν υπάρξει κάποια αλλαγή στην κυβέρνηση ε, στις ε, χώρες αυτές και αλλάξει η πολιτική τους και κάποιες χώρες αλλάξουν στάση και έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν ενώ προηγουμένως δεν συμμετείχαν. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι οι δύο συμβαστικές τροπολογίες που έχουν να κάνουν με αυτό το θέμα είναι η C και η H. Παραμένει ανοιχτό πάντως για τις χώρες μέλη το κατά πόσο θέλουν ή όχι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το Ταμείο όμως θα υπάρχει στη διάθεση των απόρων. Θα ξέρετε επίσης ότι η Επιτροπή μας έχει εκφράσει την άποψη ότι τα 2,5 δισεκατομμύρια δεν φτάνουν για το ταμείο αυτό, γιατί είναι λιγότερα από το σημερινό MDP, παρόλο που έχει πιο περιορισμένο στόχο. Ω αρμόδια επί τη ουσία επιτροπή, εμεί αλλά και άλλε επιτροπέ και επιτροπή ελέγχου προπολογισμών κλπ. έχουν προτείνει η χρηματοδότηση να παραμείνει σε επίπεδο MDP, δηλαδή 3,5 δισεκατομμύρια. Εμείς θέλουμε να προτείνουμε στην έκθεση που θα εγκρίνει η Επιτροπή μας να αναφέρονται τα 3,5 δισεκατομμύρια, να αναφέρεται το ποσό δηλαδή, αυτό θέλουμε, να αναφέρονται τα 3,5 δισεκατομμύρια. Άλλες ομάδες πιστεύουν ότι είναι καλύτερα ε, να αφήσουμε περιθώριο για κάποια διαπραγμάτευση του ποσού σε κάποιο μετέπειτα στάδιο. Άρα θα υπάρχουν δύο διαφορετικές τροπολογίες για το θέμα αυτό. Η θέση μου πάντως είναι να αναφέρετε το ποσό στην έκθεση και να μπορέσουμε να πετύχουμε τη χρηματοδότηση των 3,5 δισεκατομμυρίων. Και όσον αφορά τώρα την πλατφόρμα διάδοσης, εδώ υπάρχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά την ε, online διάδοση των πρακτικών που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα και πώς θα λειτουργήσει αυτό. Υπάρχουν προτάσεις για ιστοσελίδες, Υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές διατύπωσης πιο πολύ από τις άλλες ομάδες. Τέλος, θέλω να πω ότι όσον αφορά την ψηφοφορία των τροπολογιών όταν ψηφίσουμε. Εάν η θέση των σοσιαλιστών είναι αποδεκτή και η μνήα στην συμμετοχή των κρατών μελών αφαιρεθεί ή αν αντίθετα οι τροπολογίες των άλλων πολιτικών ομάδων υπερψηφιστούν το συμβαστικό κείμενο θα παραμείνει. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Να ξέρετε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά για την έκθεση αυτή. Και έχουμε βελτιώσει κατά πολύ το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπήρξε πολύ καλή επίσης συνεργασία μεταξύ των σκιωδών εισηγητών από τις 34 συμβαστικές τροπολογίες να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές πάρα πολύ καλές. Δύο είναι βασικά τα ζητήματα, τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Αυτά προς το παρόν και περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν, πριν δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους, Έχουμε κάποια θέματα νομική βάση για το κείμενο αυτό, αλλά πριν να συζητήσουμε αυτό, να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Κομισιόν, την κυρία Γκουίνεφ. Ε, thank you very much. Ε, Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς πράγματι Θέλουμε να συμπενθυμίσουμε τη θέση της Κομισιόν, η οποία έχει ε, καταθέσει μια πρόταση σχετικά με ένα εργαλείο για να βοηθηθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, που αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια. Έχουμε λοιπόν ε, κυρίως παιδιά που υποφέρουν από ακραίες στερήσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει και μια τεχνικής φύσεως παρατήρηση. Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι οποιοδήποτε εθελοντικό σύστημα με την έννοια ότι μπορεί να περιλαμβάνει την ε, καταγραφή από πλευράς ε, κράτους μέλους ή και την κοινοποίηση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ε, ε, διανομή τροφίμων. Ε, αυτό αφορά την ε, περίοδο 13-14. Η ΜΚΟ δέχεται κατά την περίοδο αυτή να αντιμετωπίσουν κάποιες αναταράξεις στην διανομή των τροφίμων. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους. Ο κύριος Όρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, να σας πω ότι δεν χάρηκα πάρα πολύ που σήμερα δεν ψηφίσαμε την έκθεση αυτή. Βέβαια δεχόμαστε αυτή την αναβολή, αλλά σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά στοιχεία, ναι, φυσικά μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Όμως, Ταυτόχρονα θα έχουμε και κάποιο περιθώριο ελιγμών. Βεβαίως, ε, σεβόμαστε απόλυτα την απόφαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, ακούσια ή την υποχρεωτική συμμετοχή, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο αυτό το θέμα. Δεν αρκεί να πούμε ότι α, ένα κράτος μέλος θέλει να συμμετάσχει και ένα άλλο όχι. Δεν αρκεί αυτό. Όταν ε, μιλάμε για ευρωπαϊκά προγράμματα ε, επιστηστικής βοήθειας ε, δημιουργούμε ένα άλλο ταμείο και πώς το κάνουμε αυτό θέτοντας σε τέλος ένα εφισταμένο πρόγραμμα και μάλιστα με λιγότερα κονδύλια και έτσι λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν λιγότεροι ενδυνάμοι δικαιούχοι και δυστυχώς θα αλλάξει η κατάσταση αν υιοθετήσουμε αυτή την προσέγγιση. Δηλαδή τώρα θα πρέπει να επιλύσουμε το πρόβλημα ε, με λιγότερα χρήματα. Ενώ η... το όλο εγχείρημα γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο. Υπάρχει μια προσέγγιση που λέει να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αυτό θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο τις αποφάσεις που λαμβάνονται στους κόλπους του Συμβουλίου και η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο πολύπλοκη. Δεν είναι τυχαίο το ότι η συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα είναι τόσο οξία στο Συμβούλιο. Νομίζω πως ε, σε ό,τι αφορά στο θέμα της νομικής βάσης και στο θέμα της κοινοποίηση. Μπορούμε να βρούμε λύσεις, αλλά πριν τις 20 Μαΐου, πριν την τελική ψηφοφορία, θα επανέλθουμε στο ΕΛΚ, στη συζήτηση όλων των πιθανών λύσεων. Όμως, ας μην αμφισβητούμε το ότι υπάρχει καλή βούληση σχετικά με την εκούσια, την υποχρεωτική συμμετοχή. Απλώς είναι πολύπλοκη κατάσταση. Τώρα, ας μιλήσουμε για την πλατφόρμα. Δημιουργούμε ένα ταμείο. Φυσικά θα έχουμε λιγότερα κονδύλια, όμως για μια ακόμη φορά δημιουργούμε νέες δομές, όπως είναι αυτή η πλατφόρμα διάδοσης. Έτσι λοιπόν, τι Δημιουργούμε όλο ένα και περισσότερες πλατφόρμες και δομές, ενώ έχουμε όλο ένα και λιγότερα χρήματα να δαπανίσουμε για τους απόρους. κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να έχουμε μία επιγραμμική λύση, μία λύση στο ίντερνετ, για να μην ξοδεύουμε χρήματα για μετακινήσεις ε, ή για συνεδρίασεις. Ε, όμως, ποιος είναι ο στόχος μας. Είμαστε ανοιχτοί για οποιοδήποτε συμβεσμό, όμως θέλουμε να δαπανίσει λιγότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις δομές, αλλά ε, προκειμένου να δαπανίσει περισσότερα για όσους έχουν ανάγκη. Για τους απόρους δηλαδή. Αυτό είναι ο στόχος μας. Ανεξάρτητα με το ότι είμαστε ανοιχτοί για την εξέβρεση συμβιβασμού και Φυσικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταβάλουμε περαιτέρω προσπάθειες ε, για να καταλήξουμε σε αυτό το συμβιβασμό πριν να πάμε στη συζήτηση με το Συμβούλιο. Αλλά ανεξάρτητα με τη δική μας στάση απέναντι στο συμβιβασμό, εγώ πάρα πολλές φορές ήδη έχω τονίσει ότι με αυτή τη νέα λύση, με αυτό το νέο ταμείο, θα έχουμε τελικά λιγότερα χρήματα στη διάθεσή μας και θα έχουμε λιγότερους δικαιούχους. Επομένως είναι σοβαρή η κατάσταση. Και μάλιστα αναρωτιόμαστε αν θα είναι δυνατόν να λειτουργήσουν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ από την πλευρά του ΕΛΚ. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάθε δυνατή λύση πριν από την ψηφοφορία στις 20 Μαΐου. Ε, να ζητούμε λοιπόν το συμβιβασμό και τις λύσεις. Ή... Το πνεύμα ήταν συμβαστικό στις συνεδριάσεις ε, που υλοποιήθηκαν και σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Πριν να συνεχίσουμε με τον κατάλογο των ομιλητών, εγώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι ενίοτε στην Επιτροπή μας, που είναι μάλιστα Επιτροπή Περιγνωμόνων, για τα θέματα αυτά υπάρχει μια αμφισημία για το από πού θα έρθουν τα χρήματα για το Ταμείο Απόρων. Και νομίζω ότι συνεχίζεται να υπάρχει αυτή η σύγχυση ότι τα χρήματα που δεν θα χρησιμοποιούνταν για το Ταμείο για τους απόρους θα ήταν διαθέσιμα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σαν να υπήρχαν συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ των δύο. Καταλάω ότι ορισμένοι συνάδελφοι λένε όμως εμείς δεν ε, θεωρούμε ως προτεραιότητα το Ταμείο Ενίσχυσης των Απόρων, η πραγματική μας προτεραιότητα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έτσι λοιπόν αν έχουμε μια εκούσια βάση θα μπορούμε να έχουμε τελικά περισσότερα χρήματα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, γιατί δεν θα διαθέσουμε τόσο για το Ταμείο Πόρων. Όμω, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το είπαν ξεκάθαρα. Και ακολουθούν ακριβώ την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Γιατί η νομική βάση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι η εξή. Θέλει να βοηθήσει την απασχόληση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Έτσι λοιπόν, αν πούμε ότι τα χρήματα από το Ταμείο Ενίσχυση των Απόρων μπορούν να πάνε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Αμέσω ανοίγουμε τη δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο όπου κάποια κράτη-μέλη θα πούν όμως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ε, βοήθεια για την ανάπτυξη έτσι λοιπόν όσοι λένε να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να δαπανίσουν ε, τα χρήματα είτε στο ένα ταμείο είτε στο άλλο, μπαίνουμε σε μία παγίδα, σε μία πραγματικά δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή προτείνοντας ένα ακούσιο πρόγραμμα αφήνουμε την επιλογή στα κράτη. Προτείνοντας ένα ακούσιο πρόγραμμα πραγματικά παίρνουμε το ρίσκο να κλείσουμε αυτή τη διέξοδο που έχουμε και να επιτρέψουμε στο Ταμείο Ενίσχυση των Απόρων να υλοποιηθεί. Η κυρία Κορνελίσσεν και κατόπιν η κυρία Μωρήν Σαρτιέ. Um, I think we need to find... Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να βρούμε κάποια λύση για αυτό το θέμα και να εξασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον όλα αυτά τα χρήματα ε, θα χρησιμοποιούνται για κοινωνικούς σκοπούς ε, και δεν θα επιστρέψουν πίσω ε, στον κοινωτικό προβλήσμα. Αυτό πρέπει να είναι το οδηγονήμα για μας και δεν θα πρέπει να επιστρέφουν στο χρηματοπιστωτικό ταμείο. Νομίζω ότι υπάρχει παρεξήγηση και ανάμεσα στις ΜΚΟ και από πλευράς κοινωνίας ότι δεν πρόκειται για φρέσκα χρήματα, ότι εντάσσονται και αυτά στα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων. Τώρα βέβαια έχουμε κάποιο χρόνο μπροστά μας ε, για να συζητήσουμε. Το έχουμε συζητήσει διαμακρών με τους σκιοδησηγητές ε, και με την Επιτροπή για τους πράσινους. Το βασικότερο είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από το τρέχον ε, σύστημα, από το 2014 και μετά δεν θα πεινάσουν ή ούτε και θα έχουν και λιγότερα στη διάθεσή τους. Να διασφαλίσουμε ότι τα περισσότερα χρήματα θα πάνε στους φτωχότερους ε, στα περισσότερα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να υπάρξει είναι ότι το ταμείο αυτό θα πρέπει να είναι προαιρετικό. Γιατί οτιδήποτε άλλο απλά δείχνει έλλειψη αλληλεγγύης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 19 χώρε ε, που χρησιμοποιούν 500 εκατομμύρια το χρόνο και αυτέ είναι πραγματικά οι φτωχότερε ε, χώρε αν τώρα καταλήξει το, καταλήξουν στο 2,5 δις, ε, το ποσό θα μειωθεί και αν διαιρεθεί για το 27 αντί για το 19, ε, δεν χρειάζεται να είναι κανείς ε, αυθεντία στα μαθηματικά για να διαπιστώσει ότι τα χρήματα θα είναι λιγότερα στις φτωχότερες ε, χώρες. Ακόμα και αν το 2,5 πάει στα 3,5 στο πλαίσιο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, πάλι οι περισσότερες χώρες θα πάρουν λιγότερα χρήματα γιατί θα αποφεληθούν και χώρες όπως ε, η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία. Στη δική μου τη χώρα, α πούμε, η, ε, την Ολλανδία, η κυβέρνηση είναι σε θέση να διασφαλίσει ε, διατροφή για όλους τους πολίτες ε, αν έκανε τις σωστέ επιλογές. Αλλά οι άποροι στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες δεν είναι τόσο τυχεροί. Εξαρτώνται από εμά αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν κάτι να στηριχθούν εάν τώρα εμεί αποσύρουμε τη χρηματοδότηση. των παραμείνει η χρηματοδότηση ε, κατ' ουσίαν ε, υποχρεωτική. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε τα τρόφιμα από τους στοχούς Έλληνες και Ουγγρούς ε, και τα δίνουμε σε άλλους Γερμανούς που δεν τα ανάγκη και αυτό δεν είναι αλληλεγγύη. Πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποια λύση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια τροπολογία για τα ε, κριτήρια κατανομής ε, και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το τρέχον πρόγραμμα για ε, τα τρόφιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι ας πούμε η Τράπεζα Τροφίμων στην Ουγγαρία δεν θα περιορίσει κατά το ίμιση τα τρόφιμα που διαθέτει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτήν ε, θα βασίζεται η τράπεζα περισσότερο στην πραγματικότητα και όχι τόσο στα στοιχεία της Eurostat. Η τελευταία μου παρατήρηση. Η Επιτροπή είπε ότι αν είναι προαιρετική η διάθεση, ενδεχομένω να υπάρξει καθυστέρηση. Και γι' αυτό το λόγο και εμεί ε, περιλαμβάνουμε μία παράγραφο που αφορά σε ε, προσωρινά μέτρα. Γνωρίζω, διαδικαστικά αυτά όλα είναι δύσκολα, αλλά επίσης γνωρίζω ότι όταν υπάρχει βούληση βρίσκεται τελικά μια λύση. Μια λύση για να βοηθηθούν οι άποροι όσοι έχουν ανάγκη, οι 19 αυτές χώρες που το χρειάζονται μέχρι να υπάρξει ε, το επόμενο πρόγραμμα. Ε, το πώς ε, αντιμετωπίζουμε την αλληλεγγύη, αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από μία μικρή καθυστέρηση και ίσως η πρόταση να έπρεπε να έχει κατατεθεί και λιγάκι νωρίτερα η κυρία Μωρήν Σαρτιά και κατόπιν η κυρία Καρυμαντελή. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που μπορούμε να συζητήσουμε ένα τέτοιο θέμα όπως αυτό και να εκφράσει ο καθένας τις ιδέες του. Για μένα είναι πολύ απλό για το θέμα του Ταμείου για τους Απόρους. Νομίζω ότι είναι η πολιτική Ευρώπη και το πώς αντιλαμβάνονται οι συμπολίτε μα στην Ευρώπη, θέματα που διακυβεύονται εδώ. Δηλαδή, μιλάμε για οικονομική αλληλεγγύη και αυτό το Ταμείο Βοήθεια στους Απόρους θα πρέπει να μας επιτρέψει να θέσουμε σε εφαρμογή την κοινωνική αλληλεγγύη της Ευρώπης προς το σύνολο των συμπολιτών μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι θεμελιώδες και θα πρέπει να επαγρυπνούμε, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το θέμα αυτό, γιατί ε, οι ευρωεκλογέ απέχουν ένα μόλις χρόνο και με την κρίση που εξακολουθούμε να βιώνουμε είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα αυτό και οι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας από όλες τις χώρες ε, βλέπουν ε, πώς η Ευρώπη μπορεί να προσφέρει βοήθεια στους απόρους και εγώ προσωπικά πιστεύω πως αυτή η πολιτική επιλογή της κοινωνικής ε, αλληλεγγύης είναι σημαντική, την προσυπογράφω απολύτως και επομένως ε, πιστεύω πως αυτή η βοήθεια θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ε, που υποφέρουν γιατί δεν θα ήθελα να στιγματίσουμε την ταδίτη την χώρα σήμερα Άκουσα όλα όσα υπόθηκαν και είναι πάντοτε ίδιες χώρες που κατονομάζονται, που τις δεκτυλοδείχνουμε και υπάρχουν άλλες χώρες που μπαίνουν στην, ε, ε, ως προτεραιότητα σαν να μην υπήρχαν φτωχοί παντού όμως εγώ μπορώ να σας πω ότι η φτώχεια δεν έχει σύνορα ούτε και η βοήθεια στους απόρους έχει σύνορα πρόκειται για μια ευρωπαϊκή αξία αλληλεγγύης και πρέπει εδώ να τη θέσουμε σε εφαρμογή. Και κάτι δεύτερο, Πρόεδρε, στη συζήτηση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με το να παρουσιάσουμε το ποσό του ταμείου. Τώρα αυτό το χι, ακόμη και αν είναι τέσσερα δεν μου αρέσει. Θα προτιμούσα και πρότεινα μια τέτοια τροπολογία να βάλουμε αυτά τα τρία δις, 3,5 δις που θέλαμε για αυτό το ταμείο. Διατηρούμε το αντίστοιχο αυτού που είχαμε διαπραγματευτεί πριν από την κρίση και για την περίοδο 2007-2013. Και δεν μπορείτε να με κάνετε να πιστέψω ότι αν βάλουμε αυτά τα χιχιχι θα μπορέσουμε να έχουμε πάνω από 3,5 δις. Εγώ αυτό που θέλω είναι ότι αν βάλουμε 3,5 δις, ε, θεωρώ ότι εγγυόμαστε αυτό το στόχο αλληλεγγύης, κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό ήταν το δεύτερο σχολείο μου. Νομίζω ότι πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Και στη συνέχεια και βάσει και όσων είπα στην ανάλυση μου, κατανοείτε ότι εγώ θα ήθελα να είναι ανοιχτή σε όλους η συμμετοχή. Φανταστείτε αύριο να είστε σε μια κυβέρνηση, σε μια από τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν θα είχε εγγραφεί στην αρχή σε αυτή τη συμμετοχή ε, στο Ταμείο για τη βοήθεια στην απόρριση και θα αναγκαστείτε να πάρετε την απόφαση να ε, μειώσετε ε, την ε, βοήθεια αυτής της απόρρωσης και καταλαβαίνετε τι αρνητικ, πόσο αρνητικός θα είναι ο αντίκτυπος και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι σε μια τέτοια κυβέρνηση για πολλούς λόγους. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν πολύ πιο δίκαιο να προβλέψουμε την πρόσβαση σε ευρύ επίπεδο και Στη συνέχεια τα κράτη να οργανώσουν τη βοήθειά τους όπως επιθυμούν. Πιστεύω πάντως ε, σε κάθε περίπτωση ότι βρισκόμαστε στην έναρξη των συζητήσεων γιατί βλέπουμε ότι στο ιστορικό πολιτικών ομάδων ε, υπάρχουν αποκλίνουσες θέσεις, μπορούμε να έχουμε διάφορες εθνικές θέσεις αλλά σε ό,τι με αφορά, Πρόεδρε, αυτή τη γραμμή θα υπερασπίσω. Ευχαριστώ η κυρία Ντέλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ευθύνη για τη συμμετοχή αυτή. Γιατί αν μας λένε ότι μεθαύριο θα είναι σε θελατική βάση και θα υπάρχει καθυστέρηση, ε, καθυστέρηση ξέρουμε μπορεί να είναι έξι μήνες και ένας χρόνος εδώ στην Ευρώπη. Αν λοιπόν περιμένουμε έξι μήνες ένα χρόνο, καταλαβαίνετε ότι οι άποροι δεν θα παίρνουν τίποτα. Ε, όχι λοιπόν. Η θέληση αυτή πρέπει να φαίνεται και να αντικατοπτρίζεται στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ότι όλοι μαζί θα προχωράμε. Το να μου λένε σε θελοντική βάση δεν θα χρησιμοποιούμε τα κονδύλια, το ταμείο αυτό, όχι δεν πρόκειται μόνο για την επισητιστική βοήθεια, πρόκειται για τους απορούς. Έχει να κάνει με τη φτώχεια που πλήττει και τους άστεγους και τα παιδιά. Αν λοιπόν κάποιο μπορεί να μου αποδείξει ότι από του 27 υπάρχει κάποια χώρα που δεν έχει άπορους, που δεν έχει φτωχά παιδιά, εντάξει, τότε να είναι σε θελοντική βάση. Σήμερα όμως η υποχρέωση τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πια στους δρόμους ζητιάνους. Λοιπόν, η Επιτροπή Προπολογισμών έχει ήδη ε, ψηφίσει για την επιστημιστική βοήθεια. 3,5 δεν μπορεί λοιπόν εμείς να βάλουμε στην εκθεσή μας ε, χι, χι, χι. Όχι. Πρέπει να υπάρχει ποσό. Όπως έγινε και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τουλάχιστον τα 3,5 δις. Χρειάζεται κάποιο συντονισμό τέλος πάντων. Τρίτον. Θέλω να επανέλθω σε κάτι το οποίο δεν ε, συζητήσαμε καθόλου, την απλοποίηση των διαδικασιών. Και εδώ πρέπει να κάνουμε κάτι, ώστε το νέο αυτό ταμείο μεθαύριο να μπορέσει πραγματικά να λειτουργήσει. Για αυτό το θέμα λοιπόν της απλοποίησης των διαδικασιών πρέπει επίσης να συζητήσουμε και να κάνουμε κάτι. Τώρα για τις διαφορές με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Για μένα είναι σαφές. Όταν στην Επιτροπή μας αυτή βάλαμε μια πλατφόρμα για τον αγώνα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, είχαμε πει τουλάχιστον 20-25% του κοινωνικού ταμείου για το πρόγραμμα αυτό. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το Ταμείο Βοήθειας. Το Ταμείο Βοήθειας είναι να βοηθήσουμε στις επίγουσες καταστάσεις τους άπορους, ενώ το κοινωνικό ταμείο ασχολείται με την ένταξη, με, τη... με διάφορα αλλά πιο μακροπρόθεσμα ζητήματα. Ενώ το Ταμείο αυτό βοήθειας είναι βραχυπρόθεσμα. Το κοινωνικό είναι ένα όραμα για αργότερα, για το μακροπρόθεσμο. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, είναι και το ένα και το άλλο. Μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε τους άπορους και μετά το κοινωνικό ταμείο θα φροντίσει για να ενταχθούν στην κοινωνία και πάλι. Αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να αγωνιστούμε στις συζητήσεις. Και δεν τελειώνω με αυτό. Υπάρχει και ένα συμβιβασμός, ο οποίος δυστυχώς αποκλεί την δυνατότητα συμμετοχής. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, κυρίως για τα διάφορα κοινωνικά μπακάλικα και άλλες τέτοιες δομές. Εγώ θέλω πραγματικά αυτά τα αλληλέγγυα και κοινωνικά μαγαζιά να ληφθούν υπόψη και να συζητήσουμε για το πώς θα μπορέσουν και αυτά να υποφεληθούν από το Ταμείο. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για χώρους διανομής της βοήθειας. Και το υπογραμμίζω αυτό. Δεν πρόκειται μόνο για την διανομή. Πρόκειται για μια ολόκληρη διαφορετική σύλληψη που αναπτύσσεται. Και πρόκειται και για χώρους που γίνονται συζητήσεις και ανταλλαγές. Αυτά. Ελπίζω λοιπόν και αυτό το ζήτημα να συμπεριληφθεί μέσα σε ένα μελλοντικό συμβιβασμό που θα κάνουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ η Μαριάν Χάρκιν και μετά ο Αλεξάνδρο Σέρκας. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, έγιναν πολλά σχόλια από διάφορα μέλη. Εγώ θέλω να πω ότι η συγκήτριά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί συνεργαστήκαμε εξάλλου και πολύ καλά την ευχαριστώ για την προσπάθειά της προφανώς ακόμα υπολείπονται αρκετά ανέφερα όμως τρία θέματα ε, τη συμμετοχή και την διανομή νομίζω ότι το βασικότερο εδώ είναι να δούμε κατά πόσο όλα αυτά θα είναι προαιρετικά ή ε, δεσμευτικά και εδώ πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετά θέματα ένα πράγμα που με απασχολεί είναι αυτή η μικρή ε, πλειοψηφία που μπλοκάρει στο Συμβούλιο. Έχω μιλήσει με κάποιους ε, συναδέλφους ε, και έχω αποκτήσει απαντήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, ας πούμε, έχουμε το δικό μας σύστημα που λειτουργεί καλά. Δεν θέλουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα, λένε, που να μας το επιβάλλουν. Ίσως να είναι αυτό σωστό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω και ποια είναι η άποψη των υπολείπων κρατών μελών. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στις ε, συζητήσεις μας. Άκουσα το τι είπαν οι συνάδελφοι σχετικά με την κοινωνική αλληλεγγύη, ότι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή όλοι οι πολίτες και ορισμένοι ε, μάλλον ότι όλοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ίδιους όρους σε όλα τα κράτη-μέλη. Πάντως εδώ υπάρχει ένα δίλημα και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε τη λύση στο δίλημα. Επίσης συζητάμε για το από πού προέρχονται τα χρήματα ε, αν θα έχουμε το 2,5 δις ή τα 3,5 δις, νομίζω οι περισσότεροι κατανοούν ότι τα 2,5 ε, δις ε, δεν αρκούν. Βεβαίως η δική μου η ομάδα θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να αυξήσουμε γραμμές στον προϋπολογισμό. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς εχθέ, αλλά μάλλον την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη θα επιτευχθεί ε, συμφωνία. Έχουμε λοιπόν συζητήσει διαμακρών με την Κομισιόν για αυτά τα θέματα και πολλοί από εμάς ε, έχουν θέσει την ερώτηση κατά πόσον είναι δυνατόν ε, χρήματα που δεν έχουν δαπανηθεί να επανέλθουν στον κοινοτικό προπολογισμό. Αν θυμάμαι καλά, η απάντηση τη Κομισιόν είναι ότι όλα μπορούν να γίνουν. Και ε, τέλος, ε, δεν νομίζω ότι φωτιστήκαμε καθόλου πέρα από το ότι όλα μπορούν να συμβούν. Ίσως αυτό το όλα μπορεί να το ξεκαθαρίσει η Κομισιόν, γιατί μιλάμε για τη διαφορά από 2,5 μέχρι 3,5 δις. Αυτό το ένα επιπλέον δις από πού θα έρθει. Ε, θα περιοριστεί ένα ταμείο κατά ένα δις. Μήπως μπορείτε λιγάκι να μας το διευκρινίσετε αυτό, γιατί εμένα με ενδιαφέρει. Ο κύριος Ορί είπε ότι η ομάδα του θα συζητήσει το θέμα, βεβαίως και η δική μας. Ξέρετε, αν τελικά μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία επί του θέματος. Νομίζω αυτό θα ήταν ιδιαίτερα θετικό. Πάντως εξακολουθούν να υπάρχουν θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν, κυρίως ε, με τη βοήθεια ορισμένων κρατών μελών. Γιατί υπάρχουν μερικοί που λένε ότι δεν θέλουν να εμπλακούν σε αυτό το ταμείο. Ανέφερα λοιπόν τον προπολογισμό και την ε, πλατφόρμα διανομής. Κοιτάξτε, επ' αυτής, ε, εγώ είμαι ευτυχής που μπορώ να συνεργαστώ σε αυτό το θέμα όσον αφορά την κοινωνική καινοτομία είναι σημαντική και μπορούμε να την αναφέρουμε και εδώ. Και συμφωνώ και με τον κύριο Όρη ότι είναι σημαντικό ε, το θέμα του κόστους. Ε, αυτό το ταμείο είναι καθοριστικής ε, σημασίας για ανταλλαγή εμπειριών. Έτσι λοιπόν μια online πλατφόρμα είναι χρήσιμη. Πιστεύω πάντως ότι το βασικότερο θέμα σχετικά με το ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν επιθυμούν να εμπλακούν ε, σε σχέση με την Ολυμπιακή ε, κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτό είναι αυτό που συζητάμε εδώ και προσβλέπω σε περαιτέρω συζητήσεις με την εισηγήτρια και με τους σκιώδεις. Ευχαριστώ, Αλεξάνδρο Θέρκας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Χάρκιν έχει δίκιο. Το βασικό θέμα είναι ακριβώς το θέμα της εθελοντικής ή όχι βάσης. Λέει η κυρία Χάρκιν ότι υπάρχουν χώρες που δεν θέλουν να συμμετάσχουν. Εγώ προσθέτω ότι από αυτές που δεν θέλουν να συμμετάσχουν είναι για να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά για κάτι άλλο. Διότι με την έννοια αυτή της εθελοντικής βάσης, έτσι φτάνουμε και στην συμβαστική γάμα, C, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι αντιβαίνει στην έννοια της αλληλεγγύης. Δεν είναι όπως μας το είπε η κυρία Κορνέλισον. Δεν είναι ότι πολύ καλά υπάρχουν χώρες που έχουν λύσει το πρόβλημα, οπότε αυτές οι χώρες θα μπορέσουν να δώσουν τα χρήματα αλλού. Όχι. Η μη συμμετοχή σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσω περισσότερα αυτοί που θα συμμετέχουν. Λέει η τροπολογία ότι η συμμετοχή των χωρών θα είναι χωρίς να προκαταλαμβάνεται ότι θα πλήτεται το συνολικό ποσό. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν τα χρήματα για τους άλλους εφόσον δεν συμμετέχουν κάποιες χώρες. Μα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μιλάμε για ελευθερία συμμετοχής όταν πρόκειται για την ε, αλληλεγγύη. Εδώ τα κράτη-μέλη αυτό που θέλουν να κάνουν είναι τα χρήματα αυτά να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για κάτι άλλο και όχι για τους άπορους απαραίτητα. Μέχρι να ψηφίσουμε λοιπόν έχουμε λίγο χρόνο και νομίζω ότι οι ομάδες πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο αυτό για να αποφύγουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι να μην ε, μεροληπτούμε όταν ξέρουμε ότι απέναντί μας έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους που υποφέρουν, να μην βάλουμε τα δικά μας τα συμφέροντα πάνω από αυτά. Δεύτερον, είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι στο Συμβούλιο, άρα πρέπει να έχουμε μια ευρεία σκέψη, χωρίς να σκεφτόμαστε από ποια χώρα ερχόμαστε, αλλά ολόκληρη την κοινωνία που εκπροσωπούμε εδώ. Συνεπώς, δεν πρέπει να υπάρχει καμία συμφεροντολογική ή εθνική ερμηνεία να ακούσουμε αυτούς που δουλεύουν με τους άπορους, που δεν έχουν ε, μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους ή που δεν έχουν να φάνε. Ας ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Να δούμε αυτοί τι έχουν να μας πούν. Αυτοί πιστεύουν ότι τα χρήματα από το νέο αυτό ταμείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους κοινωνικούς λόγους, που μπορεί να είναι πάρα πολύ σωστοί και ωραίοι, αλλά είναι σαν να χρησιμοποιούμε τα χρήματα των απόρων για άλλους φτωχούς που δεν είναι άποροι ή για άλλους λόγους που μπορεί να είναι σημαντικοί λόγοι, αλλά να μην είναι για τους άπορους που δεν έχουν τίποτα. Οι ιδέες του κύριου Όρη μου φαίνονται λογικοί. Έχουμε να κάνουμε με μια τραγική κατάσταση. Ωραία το παλιό πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει επισητιστική βοήθεια για αυτούς που χρειάζονται. Έχουμε λιγότερα χρήματα ενώ χρειαζόμαστε περισσότερα για την κρίση. Ξέρουμε συνάδελφοι ότι αν ανοίξουμε την πόρτα και επιτραπεί τα χρήματα αυτά να πάνε και για άλλους λόγους πέρα από τους άπορους, τότε θα πάνε ε, για τις ανάγκες εκείνων που ήδη καλύπτονται από άλλα κονδύλια. Ας κάνουμε λοιπόν την προσπάθεια να μην σκεφτόμαστε ο καθένα τη χώρα του, ο καθένας στο κόμμα του, να σκεφτούμε τους Ευρωπαίους από όποια χώρα και αν προέρχονται. Εγώ φοβάμαι ότι αν κάποιες χώρες βάσει της αρχή της ελεύθερης διάθεσης μείνουν απ' έξω, τότε αυτό που κάνουμε είναι ότι οι Γερμανοί ε, τελικά φτωχοί θα καταλήξουν ένα αλληλέγγυο με τους Έλληνε φτωχού την αλληλεγγύη δεν τη ζητάμε ανάμεσα στους στοχούς της μιας χώρας με τους στοχούς της άλλης χώρας. Όχι. Δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ταμείο, το οποίο η αλήθεια είναι, είναι σαν ένα μωρό που είχε πολλούς εχθρούς πριν ακόμα γεννηθεί. Υπάρχουν χώρες που δεν θέλουν, για ιδεολογικούς λόγους δεν το θέλουν. Η Επιτροπή Απασχόλησης, τέλος πάντων, να μην είμαστε συνένοχοι με αυτούς που θέλουν να καταστρέψουν αυτό το σύστημα. Και όσοι θέλουν να το καταστρέψουν μιλάνε για την εθελοντική βάση, στην τροπολογία Γ, σε. Είναι όπως ο Perfectus Districtus, τον Αστερίξ, που κατέληξαν ε, τελικά να τσακώνονται μεταξύ τους. Εδώ προσπαθούν να μας κάνουν να βρεθούμε σε σύγχυση και να σπείρουν ζυζάνια διαχώνες μεταξύ μας. Όχι, είναι για τους άπορους το ταμείο αυτό, για τρόφιμα, για πράγματα τα οποία θα επιτρέψουν στους άπορους να επιβιώσουν. Και δεν με ενδιαφέρει η μία ή η άλλη χώρα. Πρέπει να είναι για όλους τους άπορους, από όπου και αν προέρχονται αυτοί. Ξαβγές, ε, Ευχαριστώ. Στην Επιτροπή αυτή φαίνεται να έχουμε μια κοινή αντίληψη ότι οι άποροι στην Ευρώπη χρειάζονται βοήθεια, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα δώσουμε τη βοήθεια αυτή. Εγώ έχω μπερδευτεί πάρα πολύ με τους όρους Complementary Fund και το Voluntary Participation με την εθελοντική συμμετοχή και το συμπληρωματικό ταμείο. Και θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις. Αν τώρα μιλάμε για συμπληρωματικό ταμείο, αυτό σημαίνει ότι αυτό το ταμείο είναι εκτός ε, του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου, θα είναι εκτός του πεδίου εφαρμογή του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Ή όπως ακούσαμε την Πρόεδρο να λέει δεν θα αποτελεί τμήμα του κοινωνικού ταμείου. Δηλαδή θα είναι εντελώς εκτός ε, του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Χρειάζομαι μια διευκρίνηση αυτό και για την ε, εκούσια συμμετοχή. Αν υπάρχουν χώρες που δεν ε, θα συμμετάσχουν, δεν θα εμπλακούν σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν ε, θα χρηματοδοτούν, αλλά δεν θα είναι και δικαιούχοι του Ταμείου αυτού. Και αν υπάρχουν χώρες που πιστεύουν ότι θα φροντίσουν οι ίδιες ε, το θέμα αυτό, θα παράσχουν οι ίδιες αυτή την επιστηστική βοήθεια, γιατί να χρηματοδοτούν αυτό το ταμείο, θέλουν ε, να ακολουθήσουν ε, εθνικά προγράμματα. Αν να θέσουν σε εφαρμογή εθνικά προγράμματα. Και κάτι ακόμη. Εγώ απογοητεύτηκα κάπως που και η Κομισιόν ε, θα ήθελε να υπάρχει και άλλου είδους υλική βοήθεια. Εγώ νομίζω ότι η επιστημιστική βοήθεια είναι η πιο σημαντική. Και ξέρουμε ότι αυτό το πρόγραμμα προέρχεται από τα γεωργικά προγράμματα. Δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί εμπλέκουμε άλλη υλική βοήθεια με αυτό το ταμείο. Και έχω κάποιες αμφιβολίες ότι μπορεί η κατάσταση να γίνει ακόμη πιο πολύπλοκη για τα κράτη-μέλη, να είναι δηλαδή πολύ δύσκολο να διαχειριστούν τα κράτη-μέλη το πρόγραμμα αυτό. Μήπως κάποιος μπορεί να μου απαντήσει αυτά τα ερωτήματα. Να μου πει δηλαδή αν είναι εκτός του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισιοκτομείου το θέμα της ακουσίας συμμετοχής. Είναι ακούσια συμμετοχή σε σχέση με το θέμα της χρηματοδότησης ε, ή του να είναι δικαιούχο το κράτο. Να διαχείρισε και σε Τζοπιάτρου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, Νομίζω όλοι γνωρίζουν λίγο πολύ τα προβλήματα. Δεν νομίζω όμως ότι βοηθάει το να λέμε ότι σε κάθε χώρα υπάρχουν ενήλικες και παιδιά που πεινάνε. Πράγματι πεινάνε. Αλλά όμως στη Γερμανία ας πούμε υπάρχουν και εκεί παιδιά που πάνε χωρίς πρωινό στο σχολείο. Αυτό όμως δεν οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν ε, οι φορείς που θα επέτρεπαν κάτι τέτοιο, οφείλεται περισσότερο στις κοινωνικές συνθήκες, στις οικογένειες κτλ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υφίσταται ένα δίκτυο και το οποίο γκαιάται ότι κανείς δεν θα πεινάει. Ε, ίσως να μην λειτουργεί αποτελεσματικά. Ναι, αλλά από την άλλη υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου δεν υπάρχουν τέτοια δίκτυα και όπου άνθρωποι πολύ συχνά πεινάνε, πεινάνε αρκετοί. Δεν έχει λοιπόν νόημα τώρα ε, να βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Τουν αντίον, εγώ ε, το βρίσκω ε, να λέει κανείς, παντού τα ίδια. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να είμαστε και λιγάκι επιφυλακτικοί όσον αφορά το προαιρετικό στοιχείο των κρατών μελών. Και κάτι άλλο, μα από πότε μπορούμε να αναγκάζουμε τα κράτη-μέλη να διεκδικούν χρήματα το να επιβάλλει κανείς ένα κράτος ε, να επενδύει αποτελεσματικά τα χρήματά του, αυτό ποτέ δεν λειτουργήσε. Άρα δηλαδή εγώ θεωρώ ότι τα χρήματα πρέπει να επενδύονται από τα κράτη-μέλη όπου πράγματι το όντι υφίσταται αναγκαιότητα. Δεσμευτικά και εξαναγκαστικά να γίνεται αυτό, νομίζω κάτι τέτοιο δεν είναι αποτελεσματικό και δεν θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε την πλειοψηφία για αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. κύριο Σπρέτο. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω το πώς ξεκίνησαν αυτές οι συζητήσεις, γιατί εγώ πιστεύω ότι από την αρχή αυτή η συζήτηση πραγματικά είναι αναξιοπρεπής, γιατί πραγματικά χρησιμεύσε για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε την καρδιά μιας κύριας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά μιλάμε για ε, ενίσχυση στους απόρους ε, γιατί έχει λάβει τέλος η ιδέα της κοινή αγροτικής πολιτικής και η ιδέα που είχαμε σε προηγούμενες θητείες ήταν ότι ακόμη και αν εξαλειφόταν αυτή η πτυχή τη κοινή γεωργική πολιτική, θα έπρεπε να συνεχίσει να υπάρχει ένα πρόγραμμα για παροχή βοήθεια στου απόρου. Αυτή η αλλαγή προ την κοινωνική πολιτική χρησιμεύει σε πάρα πολλού, είτε για εθνικά είτε ιδεολογικά συμφέροντα, ε, να προσπαθούν να ξεφορτωθούν αυτό το πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι υπάρχει βέτο από τρει-τέσσερι χώρε στο Συμβούλιο και πάρα πολλοί κρούσαμε τον κοδόνα του κινδύνου, γιατί πραγματικά μιλάμε εδώ ότι διακυβεύεται η ταυτότητα ενό πάρα πολύ σημαντικού ευρωπαϊκού προγράμματο του ευρωπαϊκού Οικοδομήματο. όταν ε, ε, ε, το βέτο να μετατραπεί σε μία ε, διατήρηση. Νομίζω ότι χάσαμε κάποια μάχη ή οπισθοχωρήσαμε από μια πολύ σημαντική κοκκίνη γραμμή για το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι ανεξήγητο. Δηλαδή πρώτα να προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το ταμείο γιατί ξέρουμε ότι έχουμε 40% ε, λιγότερα κονδύλια από αυτό που ζητούσε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχήν, θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε. Είναι ανεξήγητο κάποια στιγμή όπου όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν λένε ότι το 2020 θα έχουμε 25% περισσότερους φτωχούς σε όλα τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει 40% λιγότερα κονδύλια για να βοηθήσει τους απόρους. Εγώ νομίζω ότι είναι εντελώς αναξιοπρεπές και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να Υποστηρίζουμε τα 3,5 ε, δισεκατομμύρια. Ούτε αυτά θα αρκέσουν βέβαια να έχουμε 25% περισσότερους φτωχούς ε, τα επόμενα χρόνια. Και το θέμα του εκούσιου χαρακτήρα μου φαίνεται παράλογο γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δηλαδή εδώ μιλάμε για ένα πρόγραμμα που ούτω ή αλλω γνωρίζουμε οι φτωχοί δεν είναι του ενό κράτου μέλου ή του άλλου, βρίσκονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως σας είπα δεν είναι μια απόχρωση εδώ, δεν μιλάμε για κάτι θεμελιώδες. Αυτό το ταμείο δεν μπορεί να κρίνεται από το αν επιθυμεί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση ενό συγκεκριμένου κράτου να το εφαρμόσει ή όχι. Δεν είναι λοιπόν ένα θέμα παράπλευρο, αλλά είναι θεμελιώδε το θέμα που συζητάμε. Και δεν μπορεί ε, τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να είναι η μαγική λύση όλων των ε, προβλημάτων και όταν έχουμε κάποια διαφωνία με την Κομισιόν ή με το Συμβούλιο να τα βάζουμε όλα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει τους δικούς τους σκοπούς. Έχουμε συζητήσει το θέμα της εγγύησης για τους νόσους με το 50% που πρέπει να έρθουν από τα διευθυντικά ταμεία. Όμως δεν μπορεί να είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο που θα είναι ε, ουσιαστικά το ταμείο που θα αντιμετωπίζει όλες τις καταστροφές ε, και εκεί θα παραπέμπουμε για ε, όλα τα θέματα τα οποία διαφωνούμε. Έτσι λοιπόν αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να υπερασπίζει όταν υπερασπιζόταν πάντα. Να μην πέφτουμε σε παγίδες και όπως είπε και ο Αλεχάνδρο να συνειδητοποιούμε το εξής. Κατόπιν ε, τη συζήτηση για τον εκούσιο χαρακτήρα, πίσω από τη συζήτηση αυτή, νομίζω ότι μπορεί να κρύβεται το θέμα ε, της δυνατότητα μεταφοράς ε, του Ταμείου για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλου σκοπούς. Σήμερα, για να μιλήσουμε για τη δική μου χώρα, έχουμε 1,5 εκατομμύριο άτομα που πραγματικά τρέφονται βάσει επιστημιστικής βοήθειας και το 30% αυτών των ε, ανθρώπων δεν θα μπορούν από του χρόνου να έχουν τα μέσα για να τρέφονται καθημερινά. Έτσι λοιπόν αποτυγχάνει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά αυτή η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να επιτρέψει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, σκοπίμως έμεινα να μιλήσω στο τέλος. Ε, προέρχομαι από την Ελλάδα και συχνά πυκνά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε σε πρωτοσέλιδα μεγάλων εφημερίδων δημοσιεύματα που λένε για τα παιδιά που πεινάνε στα ελληνικά σχολεία που λιποθυμούν από την πείνα. Ε, θέλω να πω τέσσερα σημεία. Το πρώτο και βασικό σημείο είναι ότι στο επιχείρημα που άκουσα μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας να μην στιγματίσουμε τις χώρες που περνούν δύσκολα νομίζω ότι δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλοι ξέρουμε και όλες ξέρουμε ποια κράτη περνούν δυσκολίες. Απ' την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό δεν σημαίνει πως στο μέλλον κάποιες άλλες χώρες δεν θα έχουν αντίστοιχες και ανάλογες δυσκολίες. Το δεύτερο ζήτημα είναι με το ότι σήμερα σε συγκεκριμένες χώρες υπάρχουν φτωχοί, άποροι, πεινασμένοι. Όταν όμως ξεκίνησε αυτή η ιστορία από την Ελλάδα κανείς δεν είχε στο μυαλό του ότι η ίδια κατάσταση θα αρχίσει να φαίνεται να υπάρχει και σε άλλες χώρες μέλη. Το τρίτο είναι ότι οι δικαιολογίες οι οποίες προβάλλονται και με βάση τις οποίες μπορεί να καθυστερήσουμε κι άλλο, νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν μόνο αν υπάρχει πολιτική βούληση και πολιτική βούληση νομίζω ότι πρέπει, οφείλει να έχει και η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι έχει την βούληση, την πολιτική βούληση για το πρόγραμμα αυτό. Το τέταρτο σημείο είναι σε καμία περίπτωση τα χρήματα αυτά να μην μετατεθούν, να μην ξοδευτούν σε άλλους σκοπούς. Και το τελευταίο μου σημείο είναι πάρα πολύ απλό και νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι μας. Κουβεντιάζουμε πάρα πολύ, σκεπτόμαστε πάρα πολύ, αλλά εάν συνεχίσουμε να καθυστερούμε, φοβάμαι ότι οι φτωχοί και οι άποροι δεν θα έχουν τη βοήθεια τώρα που την χρειάζονται. Και την χρειάζονται αυτή τη βοήθεια τώρα αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει και με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο και με τις αποφάσεις που καλούνται να πάρουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια και πάλι, μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο για να απαντήσει ίσως την κυρία Χάρκιν. Όχι, καλώς. εισηγήτρια. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους ευρωβουλευτές για τα όσα είπαν. Ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων. όσον αφορά το πρόγραμμα FEED. Τι φάνηκε από τη συζήτηση εδώ. Φάνηκε η σημασία της αλληλεγγύης με τον κόσμο εκείνο που υποφέρει τόσο πολύ από έλλειψη τροφίμων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι είναι 120 εκατομμύρια άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια, 40 εκατομμύρια που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Και μάλιστα σε στιγμή κρίσης χωρίς προηγούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε για 2,5 δισεκατομμύρια κονδύλια για να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν ε, να βάλουν ένα πιάτο στο τραπέζι για να τέσουν τα παιδιά τους που γυρνάνε πεινασμένα από τα σχολεία γιατί ούτε και εκεί δεν μπορούν να βρουν τροφή. Άρα λοιπόν αυτή είναι η προοπτική και νομίζω ότι όλες, όλοι οι ευρωβουλευτές είπαν ότι θέλουν να δείξουν την αλληλεγγύη της Ευρώπης απέναντι σε αυτούς που την έχουν τόσο ανάγκη. Τώρα, Ήδη από την αρχή σας είπα ποια είναι τα προβλήματα. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω και εδώ, το θέμα της εθελοντικής βάσης ή όχι είναι αυτό που μένει να λυθεί. Και βέβαια, τι σημαίνει αυτή η εθελοντική υποχρεωτική συμμετοχή ακριβώς. Εδώ λέμε ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε το μερίδιο της κάθε χώρας που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους άπορους. Αυτό ακριβώς λέμε εδώ. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή τα κράτη-μέλη είτε συμμετέχουν ή όχι, αυτό θα το αποφασίσουν, αλλά πάντως όλες οι χώρες-μέλη και οι άποροι σε όλες τις χώρες θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα χρήματα αυτά. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι είναι σημαντικό, είτε υπάρχουν χώρες που μπλοκάρουν την κατάσταση στο Συμβούλιο, πρέπει να ξέρουμε ότι και εκεί μετά από μερικά χρόνια μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση. Και άρα μπορεί να αλλάξει άποψη χώρα και να θέλει να συμμετέχει μετά. Η συζήτηση πάντως ήταν σίγουρα ενδιαφέρουσα εδώ και θα δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε και να λύσουμε το θέμα αυτό της συμμετοχής. Να ξέρετε ότι είναι πρόγραμμα πάντως για τους άπορους όλων των χωρών. Αυτό είναι στοιχείο που είναι στην καρδιά του προγράμματος. Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω είναι ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε ένα πολιτικό όργανο. Και είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη στήριξή μας στο πρόγραμμα αυτό, πόσο σημαντικό το θεωρούμε και πόσο σημαντική θεωρούμε την παρετέρα ανάπτυξή του. Είναι επίσης σημαντικό το ποσό να είναι 3,5 δισεκατομμύρια και να ανεβάσουμε τον πύχη, γιατί πρέπει να έχουμε το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης στο νέο πρόγραμμα, όπως είχαμε και στο τωρινό τρέχον MDP. Κατά τα άλλα, σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή σας και όσον αφορά την ε, πλατφόρμα διάδοσης. Να ξέρετε ότι έχει να κάνει με τα χρήματα που δίνει η Επιτροπή και πουθενά δεν προτείνεται ότι η πλατφόρμα αυτή ε, θα επηρεάσει τις προπολογισμού των χωρών μελών για τους άπορους. Χαίρομαι πάντως που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την συζήτηση εκτενώς και ελπίζω ότι θα φτάσουμε σε συμπεράσματα. Προσλέπω την ψηφοφορία και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο για την στήριξη μας όσον αφορά το πρόγραμμα FEED. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Με την άδειά σας επιτρέψτε μου να επανέλθω λίγο σε αυτό που ρώτησε η κυρία Σαγιά. Διότι θέλω να σας καθισχάσω στα συμπεράσματα του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου με το CFP δεν μιλάει για διακυβερνητικό ταμείο δεν πρόκειται για ενισχυμένη συνεργασία εδώ είναι στα πλαίσια του πολιτούς δημοσιονομικού προγράμματος. Τώρα αν είναι ένα υπομέρος του κοινωνικού ταμείου και τα κράτη-μέλη να μπορούν τα χρήματα αυτά να τα βάλουν για τους άπορους ή για το, τα κοινωνικά, αν ήταν έτσι, τότε θα μπορούσε να υπάρχει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την νομική βάση του κοινωνικού ταμείου είναι για την απασχόληση και όχι για τους άπορους. Γι' αυτό, πάνω σε αυτό δουλεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι κάπως περίπλοκο. Θα έχουμε μία ειδική γραμμή για το Ταμείο για τους Άπορους, που δεν θα είναι στο Κοινωνικό Ταμείο, θα είναι από δίπλα. Θα ακολουθεί ή θα βρίσκεται πιο μπρος δεν θα είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί αν ήταν το ίδιο πράγμα, τότε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορούσε να αποφανθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τους άφορους. Τώρα, ε, για το κατά πόσο θέλουμε να είναι μόνο για την επισητιστική βοήθεια, πολλοί από εμάς το σκεφτόμαστε αυτό. Δυστυχώς, οι συνέπειες της απόφασης του δικαστηρίου οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κάτι ευρύτερο. Και αυτό ακριβώς ήταν και η συζήτηση που κάναμε εδώ, να δείξουμε ότι η, τράπεζα της, ε, ότι η τράπεζα ε, και η δουλειά της ευνοούν την κοινωνική ένταξη. Στις συμβαστικές προτάσεις της εισηγήτριας λοιπόν, η δικιά σας ανησυχία λαμβάνεται υπόψη, θα έλεγα με δύο τρόπους. Αφενός από τη διατύπωση, στην οποία έχουν συμφωνήσει όλες οι ομάδες, που λέει ότι στόχος του προγράμματος αυτού είναι και η επισητιστική βοήθεια και η η υλική βοήθεια. Και αυτό τι σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη αποφασίζουν άλλα μόνο επισητιστική βοήθεια και όχι διανομή, ξέρω εγώ, παλιών πλυντηρίων ή κάτι άλλο. Και αντίθετα όσοι θέλουν το κάνουν αυτό. Και αφετέρου υπάρχουν οι τροπολογίες που έχουμε από την Επιτροπή Γεωργίας και Προϋπολογισμών που αναφέρονται στα αγροτικά αποθέματα. Έχουμε μια νέα βάση, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αποθέματα, αλλά αν υπάρχουν αποθέματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα αυτό. Αυτή είναι η γνωμοδότηση που μας στέλνουν δηλαδή δύο αυτές επιτροπές και με την οποία συμφωνεί η συγκήτρια. Με τις οποίες συμφωνεί η συγκήτρια. Ήταν πολύ χρήσιμη λοιπόν η συζήτηση αυτή που κάναμε εδώ και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε κατά από καλές συνθήκες και να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ακόμα και για την ε, ε, μειονότητα που μπλοκάρει πολλές φορές, τη μειοψηφία συγγνώμη που μπλοκάρει τελικά και να καταφέρουμε να τα ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Και φτάνουμε στο σημείο 8. Θα δώσω το λόγο στην Ιούτα Στάινμπρουκ, την εισηγήτριά μας, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, αν έχουν προχωρήσει όχι, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή και την Κοινωνική Καινοτομία. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο τελευταίος ε, τρίλογος ε, έλαβε χώρα στις 23 Απριλίου. Στην ε, ημερήσια διάταξη είχαμε τα υποπρογράμματα Progress και θέλαμε να συζητήσουμε για το θέμα των νέων που αποτελεί μία από τις προτεραιότητες ε, αυτής της Επιτροπής. Θέλησαμε επίσης να συζητήσουμε για τις οριζόντιες υποθέσεις και για τις γενικότερες διατάξεις. Το πρόγραμμά μας όλα αυτά δεν δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Καταλήξαμε λοιπόν σε πολύ καλές ε, συμβαστικές ε, προτάσεις. Και εκείνο το οποίο διαπιστώσαμε είναι το εξής, ότι το Συμβούλιο ε, τάσεται κατά της, το άξονα των νέων. Υπήρξε και εμπόδιο στον οριζόντιο άξονα. Εδώ λοιπόν θέλουμε να αναφέρουμε ότι στο πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία εκεί βλέπουμε ένα είδος πιλωτικών προγραμμάτων για το σύνολο του Κοινοβουλίου. Ε, πρέπει να παρακολουθούμε ε, το πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις, ε, το τι θα γίνει τελικά με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Και αυτό πρέπει να σας πω είναι πρόβλημα, διότι εμείς επιθυμούμε ως Κοινοβούλιο να ασκήσουμε πολιτική επιρροή, κυρίως όσον αφορά τα πολιτή προγράμματα εργασίας. Γιατί λέμε ότι μέσα σε 8 χρόνια μπορεί να αλλάξουν οι προτεραιότητες, άρα δηλαδή θα πρέπει να μπορούν να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις. Το Συμβούλιο διαφώνησε και η Επιτροπή βέβαια και επιτρέψτε μου να κάνω και μία προσωπική παρατήρηση. Η Κομισιόν το ρόλο της ε, στον τριμερή διάλογο ε, δεν τον αξιοποίησε, δεν στάθηκε στο ύψος της. Η Κομισιόν ήταν περισσότερο ε, ένας πολιτικός μοχλός και είναι μακράν, απέχει μακράν του ευκταίου. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για μας είναι ότι το Κοινοβούλιο θα εξακολουθήσει να ασκεί επιρροή. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ε, ως ε, σκιώδεις εισηγητές ε, αναφέραμε ότι είναι πολύ σημαντικό για μας να διαφυλάξουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Κατόπιν, το Συμβούλιο διέκοψε τις διαπραγματεύσεις η πρόεδρός μας, η κυρία Περές, έστειλε μία επιστολή στο Συμβούλιο για να καταστήσει σαφή τα επιχειρήματά μας. Γιατί δηλαδή πιστεύουμε ότι η κατεξιοδότηση πράξεις είναι πολύ σημαντικές για τα πολιετή προγράμματα εργασίας. Άρα δηλαδή αιτιολογούνται οι κατεξιοδότηση πράξεις ε, και αποτελούν νόμιμη βάση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα ε, δεν υπάρχουν ακόμα απαντήσεις του Συμβουλίου. Ε, το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν η επόμενη Τρίτη. Αυτήν έχουμε προβλέψει για την συνέχιση του τριμερούς διαλόγου. Ε, ίσως εντωμεταξύ βέβαια να υπάρχουν πιο επίκαιρες πληροφορίες. Κατά τα άλλα, είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν προχωρούν οι διαπραγματεύσεις. Ε, εν πάση περιπτώσει, το ε, Κοινοβούλιο θέλει να λαμβάνεται υπόψη η βούλησή του. Και αν θυμάμαι καλά, την έκθεση αυτή την εγκρίναμε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία και οι συζητήσεις με τους ε, σκιώδεις ε, οι εισηγητές προχώρησαν πάρα πολύ καλά στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου. Το Κοινοβούλιο λοιπόν κατέληξε σε μια θέση η οποία καθιστά σαφές στο Συμβούλιο αλλά και στην Επιτροπή ότι τον δρόμο πρέπει να τον διανύσουμε μαζί. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και τους εσκιοδησηγητές για την πραγματικά εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιο το λόγο. Όχι. Πολύ ωραία. Καλό κουράγιο για την συνέχεια σας ευχόμαστε. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 9. Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με τις αρμαδιότητες του κράτου σημαίας. Εγώ είμαι η για το θέμα αυτό. Έχω καλά νέα. Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο πηγαίνουν πολύ καλά. Προδεύουμε. Και αυτό σημαίνει ότι για θέματα που φαίνονται τελείως αδύνατο να βρούμε συμφωνία, τώρα υπάρχει ένα ανοιχτό πνεύμα και μάλιστα μαζί με τους σκιώδεις ε, εισηγητής που συμμετέχουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, υπάρχει καλή συνεργασία και μπορώ να σας πω ότι κυρίως με υποστηρίζει ο κυρίος Δεμπάκερ, ο σκιώδης συζήτης. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξή του στη συζήτηση με το Συμβούλιο και έχουμε κάνει πρόοδο στο θέμα της πιστοποίησης και στο θέμα των επιθεωρήσεων. Ήταν αναγνωρισμένων οργανώσεων οργανισμών. Υπάρχει μια κυρία δυσκολία ενωπιών μας και είναι το θέμα της νομικής βάσης. Γιατί όπως θα θυμάστε, όταν ε, καθορίσαμε την ε, εντολή, την πραγματευτική εντολή για αυτό το φάκελο, είχαμε πάρει πολλές διατάξεις από την Αυτιλιακή Σύμβαση, που έχει να κάνει με τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα που θα έπρεπε να επαληθεύονται από το κράτος σημαίας. Το Συμβούλιο μας λέει ότι η οδηγία αυτή βασίστηκε στο άρθρο 101 της συνθήκης, δηλαδή νομική βάση για τις μεταφορές και επομένως δεν μπορεί να καλύψει τα κοινωνικά ζητήματα που έχουν να κάνουν ε, με το άρθρο 155. Το Συμβούλιο αρχικά θέλησε το θέμα αυτό να το συζητήσει διμερώς με την Κομισιόν και φυσικά είμαστε προσκεκλημένοι σε αυτή τη συζήτηση γιατί η δική μας νομική υπηρεσία επίσης κινητοποιήθηκε για αυτό το ζήτημα αν ε, κατορθώσουμε να έχουμε αυτή την διπλή νομική βάση, την 101 και το 155 δηλαδή, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να σημειώσουμε σχετικά γρήγορη πρόοδο για το τελευταίο μεγάλο μπλοκ που μας επομένει να συζητήσουμε και έχει να κάνει με τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα που διευκρινίζονται στη Σύμβαση ΔΟΕ. Αυτά ήθελα να σας αναφέρω κατόπιν του πρώτου τριμερούς διαλόγου που έλαβε χώρα για αυτό το θέμα. Η κυρία Χάρκη. Thank you. Um, Mr. Couldn't be here today. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεμπάκερ δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα. Μου ζήτησε λοιπόν από δύο λόγια εκ μέρους του. Και νομίζω ότι η πρόεδρος είπε τα περισσότερα. Θα είμαι σύντομη. Λέει ότι πιστεύει ότι κινούμαστε προς τη κατεύθυνση. Υπήρχαν πολλές διαφωνίες μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου πριν την αρχή των διαλόγων, αλλά κινούμαστε σταθερά και πιστεύω ότι σημειώνεται πρόοδο. Η Ιρλανδική Προεδρία και οι Κομισιόν θέλουν να κινηθούν ε, προ την κατεύθυνση του Κοινοβουλίου και το Κοινοβούλιο επίση ε, είναι δυνατόν να βρει συμβιβασμού. Υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να συζητηθούν στου επόμενου τριμερεί διαλόγου, αλλά λέει ότι υπάρχει δυνατότητα να μπορέσει να κλείσει το θέμα κατά τον επόμενο τριμερή διάλογο, γιατί είναι σημαντικό ε, να γίνει κάτι τέτοιο, καθώ θα τεθεί το καλοκαίρι σε ισχύ ισχύ η ε, θαλάσσια σύμβαση εργασίας. Και επίσης ε, λέει ότι μπορεί να βρεθεί συμβιβασμός ε, γιατί θεωρεί ότι είναι καλό το κείμενο. Μάλιστα, βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πνεύμα που διέπει αυτές τις διαπραγματεύσεις, γιατί όλοι θα θυμούνται ότι όταν είχαμε συζητήσει το θέμα της εντολής, υπήρχε σημαντική διαφωνία και όπως είπατε τώρα και εκ μέρους του σκιώδους συζητητή, οι διαπραγματεύσεις ε, γίνονται σε ένα πνεύμα καλής συνεργασίας και έχουμε και ένα διπλό στόχο στο χρονοδιάγραμμα. Θέλει η Ιρλανδική Προεδρία καταρχήν να ολοκληρωθεί το ζήτημα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, αλλά και όλα τα μέρη θέλουν να μην υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του κειμένου που έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες του κράτους λιμένα και του κειμένου που έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες του κράτους σημαία. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνουμε και αυτό το σημείο της ημερής ένταξη εδώ και θα δούμε το τελευταίο σημείο, το οποίο είναι η σύνοψη της ε, αντιπροσωπείας μας ε, στο Όσλο κατά την ε, διάρκεια της Ένωσης Ευρωπαϊκής Περιφερειακής τη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Εγώ είχα την ευθύνη για αυτές τις διαπραγματεύσεις και συμμετείχαν και ο Αλεχάνδρος Σέρκας και ο Τσαμπα Όρη. Εδώ στο κείμενο βλέπετε το κείμενο της παρέμβασής μου, όπως και το πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν δεν θα μακρηγορήσω. Απλώς ε, θα σας πω ότι είχαμε πάρα πολλές διμερείς επαφές. Σχεδόν όλες οι διμερείς επαφές που ζητήσαμε έγιναν αποδεκτές. Και μπορώ να σας πω ότι μας εξέπληξε το ότι ε, μέσα στην οργάνωση είχε σκληρύνει ο τόνος και υπάρχει μια σύγκρουση της τριμπερούς δομής με τους εκπροσώπους των εργοδοτών που θεωρούν ότι ακόμη και η βασική σύμβαση της ΔΟΕ θα μπορούσε να αναθεωρηθεί ή να επανερμηνευθεί υπό το φως της κρίσης. Και Εμείς ε, κατόπιν της ε, παρέμβασης ε, της Τρόικα, οι, ε, της Τρόικας εργοδότες θεώρησαν ότι τα όσα υπόθηκαν δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα της κρίσης. Ο Γκί Άιντερ, ο γενικός διευθυντής, επέμεινε να ενεργοποιηθεί το Κοινοβούλιο πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την επενισορρόπηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και επίσης είχαμε και κάποιες συνομιλίες με τον Επίτροπο Άντορ σχετικά με το θέμα της νομιμότητας της Τρόικας σε σχέση με τα πόσα έγιναν στην Κύπρο. Σας μεταφέρω λοιπόν το πνεύμα αυτών των ανταλλαγών, αλλά σας καλώ να διαβάσετε και το γραπτό κείμενο, τη σύνοψη είναι πολύ πιο συγκεκριμένη και λεπτομερής από όσα μπόρεσα να πω εγώ σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση. Κύριε Σέρκα, θέλετε το λόγο, όχι. Μάλιστα, υπόθηκαν όλοι. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν εδώ τις εργασίες μας ε, και θα τα ξαναπούμε στις 20 Μαΐου στο Στρασβούργο στις 7 το απόγευμα για την ε, έκτακτη συνεδρίασή μας όπου θα ψηφίσουμε ε, για το Ταμείο για τους Απόρους.